αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε την απογευματινή μα συνεδρίαση με την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Τιερή Μπρετόν. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, η έγκρισή της. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Περνάμε στην ανταλλαγή απόψε με τον Τιερή Μπρετόν και θα περάσω και εγώ στα γαλλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που δέχτηκε την πρόσκλησή μας, γιατί το νέο πράσινο σύμφωνο ε, περιέχει φιλοδοξίες όχι μόνο περιβαλλοντικού, αλλά και οικονομικού και βιομηχανικού χαρακτήρα. Και από την ικανότητά μας να μετατρέψουμε το Green Deal σε πραγματική βιομηχανική φιλοδοξία για την αγορά μας, γιατί είστε αρμόδιος και για τα ψηφιακά και για το σύνολο της οικονομίας, θα κρίνει το σύνολο της επιτυχίας του Green Deal. Αν αυτό το νέο πράσινο σύμφωνο παραμείνει μία απλώς περιβαλλοντική φιλοδοξία χωρίς να συνοδεύεται από ένα βιομηχανικό σκέλος, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας, που είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη την πρώτη ήπειρο χωρί διοξίδιο του άνθρακα, ουδέτερη από άποψη διοξίδιο του άνθρακα, το αργότερο του 2050. Οπότε έχετε μείζωνα ευθύνη, κύριε Επίτροπε, και ένα τέταρτο περίπου για να μας παρουσιάσετε λίγες εβδομάδες μετά ε, μάλλον με λίγο στο βάζει πριν ε, την επίσημη παρουσίαση της βιομηχανικής στρατηγικής που επεξεργάζεται, το συγκεκριμένο σας όραμα με προτάσεις ε, και όσο πιο απτές ε, ε, παρατηρήσεις γίνεται για, την, για θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή ΕΜΒΗ, που είναι η πιο σημαντική, όχι από πολιτική άποψη κατά ανάγκη, αλλά η πιο σημαντική από άποψη αριθμού μελών, γιατί ακόμη και μετά το Brexit θα αυξηθεί το μέγεθο τη Επιτροπής μας, τη Επιτροπής ΕΒΙ. Οπότε σημαντικό να έχουμε αυτήν την άμεση ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Έχετε το λόγο λοιπόν κύριε Επίτροπε για ένα τέταρτο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, πριν αρχίσουμε θα ήθελα να σας πω ότι Δυστυχώ έχει συντελεστεί και το Brexit, το έχουμε αφήσει πίσω μας, παρόλο που μας θλίβει ιδιαίτερος του περισσότερου. Και γενικώ σε όλη μου την επαγγελματική ζωή μιλούσα αγγλικά, εκτό από ότι όταν ήμουν υπουργό οικονομικών τη Γαλλία που μιλούσα γαλλικά. Και πιστεύω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε μετά το Brexit, έχουμε πια 4.600.000 ε, αγγλόφωνους με μητρική γλώσσα την αγγλική που παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα παραμείνει η αγγλική σημαντική γλώσσα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, ε, για να προσαρμοστώ και εγώ και να εγκαινιάσω αυτήν την εποχή μετά τον Brexit, θα μιλήσω γαλλικά. Σας άφησα λίγο χρόνο να φορέσετε τα ακουστικά σας και συνεχίζει αγγλικά ο όπως Ε, πέρασα ε, ένα μεγάλο τμήμα της ζωής μου στη Γαλλία, αλλά έχω και γνώσεις γερμανικών. Σας ευχαριστώ λοιπόν, περνάει στα γαλλικά τώρα. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας, την Επιτροπή ΕΜΒ, γιατί έχει εξαιρετικά σημαντικές αρμοδιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως ε, είπατε και εσείς, η Επίτροπος ε, και η Επιτροπή Φοντερ Λέιεν, η Πρόεδρος Φοντερ Λέιεν και η Επιτροπή έχει τη σημαντική φιλοδοξία μέχρι το 2050 να είμαστε η Ευρώπη πρώτη ήπειρος που θα επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα. Βέβαια, αυτή η φιλοδοξία θα πρέπει να υλοποιηθεί χάρη στην υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων και φυσικά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών αλλά εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σίγουρα η δική σας επιτροπή θα παίξει κέριο ρόλο. Και φυσικά ε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θέλουμε να ξαναβρούμε στην Ευρώπη ένα νέο αναπτυξιακό και οικονομικό μοντέλο που θα είναι ταυτόχρονα όμως και κοινωνικό μοντέλο. Γιατί το νέο πράσινο σύμφωνο, η νέα πράσινη συμφωνία, το New Green Deal θα συμπεριλαμβάνει και μια σημαντική βιομηχανική στρατηγική. Μια επίση τεχνολογική στρατηγική, γιατί θα κάνουμε πολλέ επενδύσει στις νέε τεχνολογίε για να τα καταφέρουμε και θα έχει και ένα σημαντικό κανονιστικό σκέλο αυτή η στρατηγική. Οπότε, αγαπητέ Πασκάλ, θα αναλάβω και εγώ όλε τι ευθύνε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου για να συμβάλλω στην υλοποίηση αυτή τη σημαντική φιλοδοξία. Άλλωστε, όπω ξέρετε, στο χαρτοφυλάκιό μου έχω και τα ψηφιακά θέματα Οπότε θα μεριμνήσω ότι και ε, η ψηφιοποίηση να συμβάλλει στην υλοποίηση της φιλοδοξίας μας και του στόχου μας. Φυσικά το σχέδιό μας είναι μακρόπνο και μακροπρόθεσμο. Θέλουμε να γίνουμε πρωτοπόροι παγκοσμίω και να πρωτοστατήσουμε στις πράσινες φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες και μέσω αυτής της φιλοδοξίας ο στόχος μας ε, θα πρέπει να είναι για τα 350 εκατομμύρια συμπολιτών μας να γίνει η Ευρώπη μια πράσινη δύναμη, μια φιλοπεριβαλλοντική οικολογική δύναμη. Και θα σας παρουσιάσω στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου μου τι μέσα θα αφιερώσουμε για να εξυπηρετήσουμε αυτό το στόχο. Έχουμε όλη επίγνωση ότι αυτή η φιλοδοξία είναι φυσικά πολύ ελπιδοφόρα, αλλά μας γεμίζει και με περηφάνεια ταυτόχρονα. Ε, αλλά ταυτόχρονα προϋποθέτει μία ρηξικέλευθη μετάβαση. Ε, και στόχος μας είναι για να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις. Και το έργο φυσικά θα είναι συλλογικό, μια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο. Και ο Φραντς Τίμερμανς έχει ως ύψιστη προτεραιότητά του αυτή τη φιλοδοξία, όπως και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως και εγώ θα συνεργαστώ με τον Φραντς Τίμερμανς, αλλά και με τον Νικόλα Σμιτ για να καλύψουμε τα θέματα κοινωνικά και ενημέρωσης και με τον Σινκεβίτσιους, ε, τον άλλο συνάδελφο επίτροπο, για να καλύψουμε όλες τις προκλήσεις. Όπως σας είπα, θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτή τη μετάβαση και επιμένω στο σημείο αυτό. Γιατί από τότε που διατυπώσαμε αυτή τη φιλοδοξία, διαρωτηθήκαμε όλοι και το συζητήσαμε και μαζί, γιατί το 2050 θέσαμε ως χρονικό ορίζοντα, γιατί είναι τα μέσα του αιώνα, όχι μόνο. Το 2050 είναι 5 συν 25, δηλαδή 5 η διάρκεια της θητείας μας για να θέσουμε τα θεμέλια για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και σε αυτό θα αφιερώσουμε όλες μας τις προσπάθειες, θα εργαστούμε νυχθημερών και 25 χρόνια, 25 χρόνια είναι μια γενιά. Και είναι μια ολόκληρη γενιά που θα πρέπει να κινητοποιηθεί για να εξασφαλίσει αυτή τη μετάβαση. Και σε επίπεδο επίρου, αλλά και την βιομηχανική μετάβαση. Η δική μου εμπειρία από τις διάφορες θέσεις που είχα στο παρελθόν, ε, γιατί ασχολήθηκα κυρίως με τη βιομηχανία, ε, έχω επίγνωση ότι για να συντελεστεί μια βιομηχανική μετάβαση χρειάζεται μια ολόκληρη γενιά και προσπάθειες μιας ολόκληρης γενιάς. Οπότε θέλουμε η μετάβαση να γίνει σε όλους τους τομείς που όλοι θα διαδραματίσουν το ρόλο τους. Και επίσης θα πρέπει να αλλάξουμε και την οτροπία μας, να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο σκέψης μας και τον τρόπο ε, των περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών πολιτικών και των μέτρων που περιλαμβάνουν γιατί τρει θα είναι οι άξονε και θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη αυτά τα τρία στοιχεία στη νέα πράσινη συμφωνία. Καταρχήν, σταδιακά θα περάσουμε από μία οικονομία περιουσία, περιουσίας, περιουσιακών στοιχείων σε μία οικονομία από οικονομία αγαθών σε οικονομία διαμοιρασμού, συνεργατική. Και επίση ε, θέλουμε μια οικονομία όχι μόνο των αγαθών αλλά και των υπηρεσιών. Και θα περάσουμε από ένα γραμμικό μοντέλο σε ένα κυκλικό μοντέλο οικονομία, στην κυκλική οικονομία. Όλα αυτά τα στοιχεία θα ληφθούν φυσικά υπόψη, όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στη βιομηχανική στρατηγική που επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και θα παρουσιάσουμε ως Θα σταθώ στα εξή σημεία. Καταρχήν, ένα σχέδιο δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που θα ανταπεξέρχεται στο ύψο των περιστάσεων και των φιλοδοξιών. Φυσικά τα κονδύλια που θα αφιερώσουμε θα πρέπει να είναι στο ύψο των φιλοδοξιών μας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει ε, την ίδρυση του Ταμείου της Δίκαιης Μετάβασης για να συμπαρασταθούμε στις πιο μειονεκτούς περιοχές που θα χρειαστούν μια επιπλέον υποστήριξη για να υλοποιήσουν αυτή τη μετάβαση. Και ήδη έγινε η σχετική ανακοίνωση που έτυχε θετική υποδοχή και από πλευρά Επιτροπή σα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όπω αναφέρθηκε στην ανακοίνωση για το νέο πράσινο σύμφωνο, μιλούμε για διόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Εδώ μιλούμε για 13 στα Αυτέ είναι οι τάξει μεγέθου στο Ταμείο Δική Μετάβαση. Οπότε θα πρέπει να κινητοποιήσουμε πολύ σημαντικά και δημόσια και ιδιωτικά κονδύλια. Και αυτό είναι ο στόχο τη φιλοδοξία μα. Και έχουμε απόλυτη επίγνωση των ποσών που χρειάζονται να συγκεντρώσουμε. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε όλα τα επίπεδα, το ευρωπαϊκό, το εθνικό, το τοπικό, το περιφερειακό. Θα πρέπει να επενδύσουμε και στις τεχνολογίες και σε βιομηχανικά οικονομικά μοντέλα που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να διασφαλίσει την ε, κυριαρχία της ε, με πράσινες οικολογικές τεχνολογίες. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ικανότητά μας ε, να ενεργοποιούμε και κρατικές συμβάσει, δημόσιε προμήθειες, που είναι ένα σημαντικό τμήμα του κοινοτικού ΑΕΠ. Και επίσης σε αυτό τα θέματα θα πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι, γιατί μερικές φορές ε, υστερούν τα κρατη Και δεν ξεκινούμε εκ του μηδενός. Ήδη η Ευρώπη ε, έχει ηγετική θέση και μιλώ κυρίως για διπλώματα ευρυσιτεχνίας. Γιατί με ενοχλεί που λέμε ότι στερούμε ή ακούω ότι στερούμε σε θέματα τεχνολογικά, ότι ε, έχουμε μείνει πίσω και στα διπλώματα ευρυσιτεχνίας. Δεν ισχύει. Και για τα πράσινα εντό εισαγωγικών. Τα οικολογικά διπλώματα ευρυστεχνία δεν το λέμε αρκετά, δεν το τονίζουμε, αλλά εμεί πρωτοστατούμε. Η Ευρώπη έχει ηγετικό ρόλο. Και έχετε περισσότερο αριθμό των πράσινων ε, διπλωμάτων ευρυστεχνία μετά την ΣΥΠΑ, Ιαπωνία και Κίνα. Και θα συνεχίσουμε να κρατήσουμε αυτό τον ηγετικό μας ρόλο σε ό,τι αφορά τα πράσινα εντό εισαγωγικών διπλώματα ευρυστέχνειας. Και αυτό είναι προ όφελο και των επιχειρήσεων όλων, ε, μικρών και μεγάλων. Επίσης θα ήθελα να σκεφτούμε πώς θα προσεγγίσουμε τις ε, αξιακές αλυσίδες στρατηγικής σημασίας, ώστε να στηρίξουμε τη μετάβαση σε όλους τους κρίκους αλυσίδας και να δώσουμε έμφαση στις τεχνολογίες που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να εξασφαλίσει αυτή τη μετάβαση. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που θα έχουμε στη διάθεσή μας και φυσικά θα και τα ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού δικαίου, αλλά όλο και περισσότερο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ε, το σχέδιο κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Τα σχέδια κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος, που το είδαμε στα πλαίσια των ε, μπαταριών ε, ή για το υδρογόνο, για παράδειγμα. Τα ευρωπαϊκά σχέδια κοινού συμφέροντος αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία και είναι ένα μέσο που θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε τακτικά. Επίσης, όπως είπε και η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε ίσως και τους κανόνες μας περί ανταγωνισμού, που θα πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του ψηφιακού κόσμου, στις γεωστρατηγικές προκλήσεις, αλλά και στις ε, φιλοδοξίες μας για το κλίμα και το περιβάλλον. Και όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να επανεξετάσουμε την πολιτική ανταγωνισμού. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Κέριο θέμα και αυτό. Και πολλοί από εσά έχετε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και σίγουρα θα με βοηθήσετε και θα γίνετε πηγή έμπνευση και για τη δική μας πρόταση. Θέλουμε πιο κυκλικό χαρακτήρα όλων των βιομηχανικών κλάδων και η οικονομία που θα εδράζεται περισσότερο στη βιωσιμότητα, στην αηφορία των προϊόντων. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Οπότε το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία ήδη είναι σε φάση εκπόνησης και θα ενταχθεί στην, στρατηγική, στην βιομηχανική μας στρατηγική. Επίσης θα επικεντρωθούμε στον κύκλο ζωή των προϊόντων, στην προμήθεια των πρώτων υλών, αλλά και στην επεξεργασία των αποβλήτων, προκειμένου να μετατραπούν τα απόβλητα και τα απορρίμματα σε ε, νέες πρώτες ύλες, γιατί ε, ε, η ανακύκλωση είναι σημαντικός τρόπος ανάκτησης δεύτερων υλών και θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε αυτή την κυριαρχία μας. Μόνο το 12% των υλικών που χρησιμοποιούμε προέρχονται από ανακύκλωση. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε αυτό το ποσοστό. Και μάλιστα 80% της ζωής ενός προϊόντος προσδιορίζεται στη φάση της, του σχεδιασμού του, της σύλληψής του. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, το τελευταίο μέτρο για τον οικολογικό σχεδιασμό μπορεί να μειώσει την ε, ενέργεια, τη χρήση ε, ενέργειας ε, κατά 150 τεραβάτ μέχρι το 2030. Νομίζω ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο μια τέτοια οικονομία για ολόκληρη την Ήπειρο. Τρίτος άξονας των μέτρων μας είναι κοινωνικές προκλήσεις και θέματα δεξιοτήτων και προσόντων. Έχω εξαιρετική συνεργασία με τον συνάδελφο Νικόλα Σμιτ και τη Γενική Διευθυνσή του. Είναι κέριο ζήτημα και θα πρέπει να είμαστε προορατικοί, να προλάβουμε τις εξέλιξεις για να... Ε, γιατί θα χρειαστούν προσαρμογές και στις δεξιότητες ε, και στα προσόντα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις πολίτες ε, για να διαφυλάξουμε το κοινωνικό μοντέλο και τις ειδικευμένε θέσεις εργασίας. Και στην βιομηχανική στρατηγική θα έχουμε ένα ολόκληρο σκέλος για τα μέτρα στήριξης ε, ε, και των δεξιοτήτων και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους πανεπιστημιακούς κύκλους. Μέχρι στιγμής έχει γίνει ήδη μεγάλη προεργασία στα θέματα αυτά και θα χρειαστεί εντατικοποίηση των προσπαθειών και σε περιφερειακό επίπεδο για να δούμε τι μέτρα στήριξη θα χρειαστούν, κυρίως οικονομικά, αλλά και ακαδημαϊκά, πανεπιστημιακά, κατάρτισης, ε, επιμόρφωσης, ε, για την ε, δημιουργία νέων, ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη, γιατί θέλουμε πραγματικά να συμμετέχουν στη μετάβαση αυτή όσο το δυνατόν περισσότεροι κλάδοι και πολίτες. Βέβαια, πολλά ερωτηματικά υπάρχουν για τη χρηματοδότηση, για τον ανταγωνισμό επίσης, γιατί αντιμετωπίζουμε δρυμή ανταγωνισμό όλες οι επιχειρήσεις και πολλές επιχειρήσεις φοβούνται ότι μήπως λόγω της περιβαλλοντικής μας φιλοδοξίας υπονομευθεί η ανταγωνιστικότητά τους λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού που θα υποστούν. Και σίγουρα θα χρειαστούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βρούμε κάποιους μηχανισμούς όπως αυτός του συνοριακού φόρου για τον άνθρακα. Και θα πρέπει να προσέχουμε ώστε τα εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες να μην προέρχονται από χώρες που έχουν ε, χειρότερες προδιαγραφές περιβαλλοντικές ή πρότυπα από εμά για να μην δημιουργηθεί αθέμετος ανταγωνισμός. Και αυτό το επισημαίνω συστηματικά στα κράτη-μέλη, γιατί είναι κέριο θέμα. Και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι ε, εσθενίζετε και εσείς αυτήν την άποψη. Να προσθέσω και άλλα δύο στοιχεία, αν μου επιτρέπετε. μιλώντας για κάποια τομεακά θέματα, πολύ σύντομα για την ψηφιακή οικονομία, για τη χημεία, για την αυτοκινηστική βιομηχανία και την βιομηχανία έντασης ενέργειας. Καταρχάς, τα ψηφιακά. Μιλούμε για ένα τομέα όλο και πιο σημαντικό, ο οποίος ε, πλαισιώνει πλέον ε, τη ζωή μας ε, απολύτως σε κάθε επίπεδο, μεταμορφώνει την δραστηριότητά μας, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που διαβάζουμε και ακούμε και βλέπουμε πλέον, ε, ε, επεξεργασία δεδομένων, όλες αυτές οι τεχνολογίες ε, αλλάζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε, που δουλεύουμε. Πρέπει λοιπόν να βελτιστοποιήσουμε την πράσινη, την οικολογική μεταμόρφωση, τροποποίηση των δραστηριοτήτων και μπορούν να συνεισφέρουν κατά 15% στη μείωση των εκπομπών που είναι στόχο μα. Επομένω πρέπει όλα αυτά να ε, είναι πιο εντατικά στην προσπάθειά μα. Εντό του τομέα αυτού πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, ε, πράσινε επιδόσεις. Σήμερα είναι πολύ σημαντικός συνεισφορέας εκπομπών ιδιαίτερα στον τομέα των δεδομένων αυτό εμείς θα το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα λοιπόν. Πρέπει να μπορέσουμε να φτάσουμε σε τεχνικές και τεχνολογίες ε, ουδέτερες ως προς τον άνθρακα. και δεν είναι καθόλου αμελητές η... Ε, το μερίδιο των εκπομπών του άνθρακα που οφείλονται στις τεχνολογίες αυτές. Επαναλαμβάνω. Και επομένως για να φτάσουμε να ε, είμαστε ουδέτεροι μια μέρα θα πρέπει να ηγηθούμε και σε αυτές τις ε, προσπάθειες, δηλαδή στο να βρούμε νέες τεχνολογίες που να είναι πιο οικολογικές. Και πρέπει και οι συμπολίτε μα να αντιλαμβάνονται και να γνωρίζουν και να του το λέμε ότι όλα αυτά τα κινητά που χρησιμοποιούμε και οι ευφυεί συσκευέ κτλ. συνεισφέρουν σε εκπομπέ. Να κάνω και μια εστίαση στη χημία αν μου επιτρέπετε, που είναι σημαντικό τομέα επίση, ε, σημαντική βιομηχανία, απαραίτητα προϊόντα, απαραίτητα και στι ε, σύγχρονε τεχνολογίε, ε, στου σωρευτέ, στι μπαταρίε και αυτό θα συνεισφέρει στην προσπάθειά μα ουδετερότητα ω προ τον άνθρακα. Εγώ δεν φοβούμαι να το πω. Έχουμε την πιο προηγμένη νομοθεσία στον κόσμο για τα χημικά προϊόντα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αερογοάς την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Κατά κινδύνων, ε, επικίνδυνων μάλλον χημικών προϊόντων, αλλά και πιο αποτελεσματική ε, ε, λειτουργίας, ε, δέσμευση ως προς όλους αυτούς τους στόχους που έχουμε θέσει στον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ε, ένα σαφέστερο πλαίσιο ώστε να έχουμε και καλύτερη συμμόρφωση και ιδιαίτερα εδώ αναφέρομαι σε πολύ σημαντικά βιοχημικά στοιχεία όπως τους ε, ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τον χημικό κλάδο να είναι υπεύθυνο, να είναι και ανταγωνιστικός αλλά και καινοτόμος για να μπορέσει και αυτός να συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου μας αλλά να έχουμε και ασφάλεια χημικών προϊόντων για τα εισαγόμενα χημικά προϊόντα. Τρίτη εστίαση πολύ σημαντική είναι τα, η αυτοκινηστική βιομηχανία. Είναι πολύ σημαντική για την οικονομία μας και την ανταγωνιστικότητά μας. Είμαστε ηγέτες εδώ, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι εδώ έχουμε πολύ πολύ ριζικές ε, διαδικασίες μεταμόρφωσης. Έχουμε δει κρίσεις και συγκεκριμένα συμπτώματα, τα γνωρίζουμε όλοι καλά, πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, να μην εγκαταλείψουμε την ηγετική μας θέση, αλλά να μην εγκαταλείψουμε και τους οικολογικούς μας στόχους. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε όλες τις επιχειρήσεις, όλες τις εταιρείε να αλλάξουν τα πρότυπα, τα μοντέλα τους και εδώ μιλούμε για μέσο μακροπρόθεσμη προσπάθεια, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε την προσπάθεια αυτή. Και θα πρέπει να συνοδεύσουμε αυτή την προσπάθεια που καλούνται να καταβάλουν οι επιχειρήσεις, διότι οι διάφορες τεχνολογικές επαναστάσεις έρχονται από το εξωτερικό και επομένως και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί να επιτηρούμε μιλώ για τα ψηφιακά στήματα, αλλά όχι και μόνο, μόνο ε, με ψηφιακά και μπαταρίες έχετε περίπου το 40% του, του, του μέσου κόστους ε, του μελλοντικού οχήματος αυτοκινήτου. Μιλούμε λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό μερίδιο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως ε, επί των δύο αυτών αξώνων γνωρίζουμε πού πρέπει να εστιαστεί η προσπάθειά μας, τώρα πρέπει αυτά να τα υλοποιήσουμε. Και αυτό είναι στόχος μας και στα πλαίσια της, του Green Deal. Εργάζομαι στο νέο πρότυπο γύρω 7 από το 2021 για να μειώσουμε τα οξύδια ε, του αζότου. Γιατί έχουμε σήμερα απαράδεκτα θα έλεγα επίπεδα ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης ε, στις πόλεις μας αυτό το νέο πρότυπο λοιπόν θα ρυθμίζει και τα πολύ μικρά σωματίδια. Μαζί φυσικά με τις εκπομπές διοξιδίου και υπόλοιπα αέρια θερμοκηπίου ε, θα ρυθμίζουμε την χρήση των μελλοντικών ηλεκτρικών οχημάτων και τη χρήση των μπαταρίων, του υδρογόνου. Ε, όλα αυτά επίσης τα, έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνεισφέρουν στο πλαίσιο αυτό και μιλώ εδώ για τις ε, μεταφορές αλλά όχι μόνο. Είναι σημαντικό επίσης οι καταναλωτές να στραφούν προς οχήματα που θα τους προσφέρονται στην αγορά που θα είναι καθαρά. Αλλά θα πρέπει να είναι καθαρά, θα πρέπει να, είναι, να διατίθενται και σε μια τιμή προσιτή. Επομένως μιλούμε για διάφορα επίπεδα και πλαίσια που αφορούν στον τομέα αυτών. Και από την 1η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουμε αυστηρή συμμόρφωση στην επιτήρηση της αγοράς για την απέτηση μη κατακαιρματισμού της αγοράς αφενός ε, και τη βούληση θέληση κάποιων κρατών μελών να προχωρήσουν πιο γρήγορα στα πλαίσια αυτά. Σα ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, αν ε, υπερεύνει το χρόνο που μου δώσατε. Είμαι έτοιμος να ακούσω τις ερωτήσεις ε, των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ. Θα γυρίσω τώρα στα αγγλικά, λέει ο Πρόεδρος. Ε, θα ακούσουμε τώρα τους ε, συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Ξεκινώντας από το ΕΛΚ, δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Είχε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο. Θα μιλήσω στα γερμανικά, όχι λόγω του Brexit, αλλά επειδή έχουμε εξαιρετικούς διερμηνείς, λέει ο ομιλητής. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τα ξεκάθαρα λόγια σας ότι προσπαθείτε να συμβιβάσετε περιβάλλον και τεχνολογία. Έχω δύο συγκεκριμένε ερωτήσει Πρώτον το θέμα των επιδοτήσεων. Το αναφέραμε παραδείγματο χάρη αν μιλάμε για παραγωγή χάλιβα ή χημικών προϊόντων χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, χρειαζόμαστε και εθνικά κονδύλια έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν να με ακούτε ε, να μιλήσω αγγλικά, αλλά τότε σταματήστε το χρονόμετρο. Δουλεύει ή όχι. Με ακούτε τώρα. Να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω και πάλι λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Σωστά είπατε ότι ο στόχος μας ε, πρέπει να είναι να συμβιβάσουμε βιομηχανία, θέσεις εργασίας ε, και προστασία του περιβάλλοντος. Έχω δύο ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στις επιδοτήσεις. Ε, θα ήθελα να μας πείτε όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Αν μια επιχείρηση, παραδείγματος χάρη, επενδύει σε παραγωγή χημικών προϊόντων ή χάλιβα χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, χρειάζεται και στήριξη από τον εθνικό προπολογισμό. Θα φροντίσετε μετά η Κομισιόν ε, να μην το θεωρήσει αυτό παράνομη επιδότηση. Δεύτερη ερώτηση αφορά το θέμα των ε, χημικών ουσιών. Έχουμε την εξή ενδιαφέρουσα κατάσταση. Και η βιομηχανία και οι περιβαλλοντικές ενώσεις θέλουν να διατηρηθεί η νομοθεσία αυτή και μετά το Brexit. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος είναι καλύτερο από την φήμη του και θεωρώ ότι η Κομισιόν σε πολλές περιπτώσεις έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Για μια φορά υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ κυκλικής οικονομίας ε, και της δυνατότητας να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατόν όλες οι βλαπτικές ουσίες, αλλά νομίζω ότι στο θέμα του διοξιδίου του χρωμίου ή του μολύβδιου στα PVC, μέχρι στιγμής η Κομισιόν έχει βρει μια λογική γραμμή, προστατεύει την υγεία και το περιβάλλον και ταυτόχρονα δεν εμποδίζει την οικονομία και δεν οθεί τις βιομηχανίες να φύγουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν όσον αφορά τον μόλιβδο και τις ε, άλλες ε, που ανέφερα τα διοξείδια του χρωμίου να διατηρηθεί. Σας ευχαριστώ Γκίτελαντ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Θα μιλήσω αγγλικά, είναι η εβδομάδα μετά το Brexit. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω και για το πράσινο deal και για το ότι θα εστιάσουμε πραγματικά στις προδιαγραφές ε, και στο μέλλον και αναφέρατε τώρα και το γύρο 7 για τα αυτοκίνητα, τον εξηλεκτρισμό. Σας ενθαρρύνω σε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα ήθελα να είστε κάπως πιο συγκεκριμένος, γιατί όταν μιλάμε για τον εξηλεκτρισμό, για τα οχήματα, πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και θεωρώ ότι οι ανάγκες θα είναι μεγάλες και να υπάρχει δυνατότητα να φορτίζει κανείς ε, το αυτοκίνητό του, αλλά ε, και τα φορτηγά στους δρόμους. Ε, πρέπει να υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα λοιπόν, να συνεργαστούμε, να συνεργαστείτε και εσείς με τους συναδέλφους σας στην Κομισιόν, έτσι ώστε η ναι, είστε αρκετά σκληρός. Ε, η άλλη ερώτηση που έχω να κάνω αφορά τι χημικές ε, ουσίε. Ε, χαίρομαι που αναφέρατε του ενδοκρινικούς διαταράκτε. Υπάρχουν όμως διαφορετικές προδιαγραφέ. Εάν δείτε τα αυτοκίνητα, τα παιχνίδια, τα καλλιτικά δεν προστατεύονται οι πολίτες της ε, Ευρώπης και εσείς πραγματικά έχετε ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια εναρμόνιση και για την εσωτερική αγορά είναι σημαντικό οι κανόνες να είναι επαρκείς, δηλαδή να μην είστε πιο αυστηροί σε έναν κλάδο από ότι σε έναν άλλον. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνουμε έτσι ώστε οι ενδοκρινικοί διαταρακτές ε, να απομακρυνθούν κάπως πιο γρήγορα γιατί το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ αργό, δεν βλέπω να προγραμματίζετε να κάνετε τίποτα μέχρι το 2023. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Για το ΡΙΝΙΟ, ο κύριος Τόρβαλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ που ήρθατε το Σάββατο που μας ε, πέρασε επισκέφτηκα το Φόστεμ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Το έργο υπάρχει εδώ στις Βρυξέλλες εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν 10-15.000 ε, νέοι που ασχολούνται με τον προγραμματισμό. Το πιο ενδιαφέρον θέμα γύρω από αυτή την υπόθεση που γίνεται στο Γαλλόφωνο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών είναι ότι δεν θα το μάντευε κανείς ότι είναι στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει θενά κανένα σήμα της Κομισιόν του Κοινοβουλίου. Τέλος πάντων, αυτοί ε, θα μας βοηθήσουν όμως γιατί έχουμε εδώ όλους αυτούς τους ανθρώπους ε, που χρειαζόμαστε τους οποίους όμως ε, θα τσιμπήσουν οι αμερικανικές εταιρείες αν δεν κάνουμε τίποτα. Ε, λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει στο GitHub 99% των έργων κινούνται με ανοιχτό λογισμικό. Έχω και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ε, και ευχαριστώ να σας βοηθήσω να έρθετε σε επαφή ε, γιατί ε, και το όνομά μου κάτι λέει σε αυτούς τους ανθρώπους. Το δεύτερο. Μιλήσατε για την αλλαγή παραδείγματος. Τις τελευταίες εβδομάδες ξαναδιαβάζω ε, το βιβλίο του Ροστόφ «Οι φάσεις οικονομικής ανάπτυξης». Γιατί, γιατί μας δείχνει ότι ε, στην αλλαγή οικονομικής ε, ανάπτυξης υπάρχουν κάποιοι κλάδοι οι οποίοι πρωτοστατούν. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποιες προσπάθειες κάνει η Κομισιόν για να μπορέσει να σχηματίσει στο κατάλληλο το άλογο. Σας ευχαριστώ. το ID παρακαλώ. Ορίλια Μπενιό. Ε, κύριε Επιτρόπε, πράγματι οι δραστηριότητε τη Επιτροπή στην εσωτερική αγορά συνδέονται με τι περιβαλλοντικέ απαιτήσει και στόχου. Σε επίπεδο περιβάλλοντο, είμαστε καταδικασμένοι να λειτουργούμε εν κενό δεδομένων ε, των ε, εισαγωγών μας και του σχεδιασμού των κωδίκων και των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να περιορίσουμε τις εισαγωγές ε, ενεργειοβόρων προϊόντων και έχουμε και εχθρούς ε, ε, του περιβάλλοντος, ορκισμένους θα έλεγε κανείς, που είναι η, τα παροχημένα συστήματα πληροφορικής. Η υποστήριξη των ευρωπαϊκών μας βιομηχανιών και επιχειρήσεων θα μπορούσε να ε, συνάδει περισσότερο με την προστασία του περιβάλλοντος. Εμείς υποστηρίζουμε τις προσπάθειες ανάπτυξης ε, κινητήρων και μηχανημάτων ουδέτερων ως προς τον άνθρακα, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να σημάνει καταστροφή της αυτοκινηστικής μας βιομηχανίας και περιορισμό των συμπολιτών μας που χρειάζονται τις μαζικές μεταφορές σε διάφορα επίπεδα. Οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις θα είναι επίσης ένα αβάσταχτο άκθος για τους συμπολίτες και τις επιχειρήσεις. Η απομάκρυνση από τον άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές επίσης που δεν αναφέρεται πουθενά και που είναι εκτός κάθε ελέγχου σήμερα. Επομένως η ιδεολογική σας τοποθέτηση είναι σαφής. Στο ρετματολόγιο που είχατε ε, κυκλοφορήσει είχατε μιλήσει κατά κάθε τάση προτεξιονισμού από πλευράς των κρατών μελών και παραθέσατε τον Ζόμονε που έλεγε ότι τα ευρωπαϊκά μας έθνη είναι πολύ μικρά για να ανταγωνιστούν με τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου, αλλά οι μεγάλες αυτές δυνάμεις είναι όλες ε, προτεξιονιστικές. Εσείς επιβαρύνετε τις εθνικές μας βιομηχανίες, τις αφήνετε ακάλυπτες στον ε, διεθνή ανταγωνισμό που ο, όπως έλεγα οι ανταγωνιστές μας είναι πρωταξιονιστές και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο φορολογικό και με ασαφείς περιβαλλοντικούς ε, στόχους. Ο κ. Ζαντό, ευχαριστώ ε, Επίτροπε. Ε, μας αναφέρετε το όρομά σας και τον στόχο σας να αλλάξετε τους κανόνες στην, στις δημόσιες προμήθειες. εργάζεστε σε ένα σχέδιο ευρωπαϊκού νομοθετήματος. Αυτό με βρίσκει σύμφωνο. Επίση, ε, περιγράψατε την κατάσταση που ισχύει για τι εκπομπέ, ε, για την ουδετερότητα άνθρακα που θέλουμε να επιτύχουμε, για τι εκπομπέ που σχετίζονται με τα ε, αυτοκίνητα, με τα πρότυπα που θα πρέπει να ενισχυθούν. Γνωρίζετε όμω ότι σήμερα αυτά τα πρότυπα, τα σκάνδαλα με το γύρο 5 και 6 συνεχίζονται. Εγώ εργάζομαι στα θέματα αυτά του διοξιδίου για τα αυτοκίνητα από το 2008 και από τότε μου έλεγαν οι παραγωγοί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο γιατί είχαν ξεκινήσει τα 4x4, ε, μετά είχαμε τα SUV και επομένως στο σκηνικό το ευρωπαϊκό ε, έχουμε ολόκληρες πόλεις που είναι έτοιμες να απαγορεύσουν ολόκληρες κατηγορίες οχημάτων όπως τα diesel. Όλα αυτά ε, συνθέτουν μία εικόνα αλλά δεν μας δίνουν προοπτική. Αν θέλετε ουδετερότητα μέχρι το 2050 ή αργότερα, θα πρέπει να φύγουμε από τους κινητήρες τους θερμικούς. Έχουμε χώρες που έχουν τοποθετηθεί για στόχους μέχρι το 2040 και που θέλουν να νομοθετήσουν για, την, για το τέλος των ε, κινητήρων ε, εσωτερικής καύσεως, των θερμικών κινητήρων, εν πάση περιπτώσει. Ο τρόπος που λειτουργεί λοιπόν η εσωτερική μας αγορά περιορίζει κάποια κράτη που θέλουν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Το σκηνικό λοιπόν αυτό της απομάκρυνσης από τους ε, παραδοσιακούς κινητήρες θα πρέπει εσείς η Επιτροπή, η ΓΑΜΑ Κλίμα αλλά όχι μόνο να μπορέσει να προσαρμόσει το νομοθετικό πλαίσιο ως προς τις κατευθύνσεις και τους στόχους αυτούς. Υπάρχει το κόνσεπτ του Pearl Harbor, όπως το έχει αναπτύξει ένας ερευνητής, πριν από το οποίο έχουμε μια ριζική αλλαγή, ένα χρονικό σημείο ριζικής αλλαγής στην αυτοκινηστική βιομηχανία, ε, το οποίο αγνοεί τα κεκτημένα των εργαζομένων, τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Επομένως, ναι, είναι ένας γενναίος στόχος αυτός που θέτεται για την απομάκρυνση από τους παραδοσιακούς κινητήρες, αλλά θα πρέπει αυτό να πλασιωθεί από την παράλληλη, ε, κατάλληλη νομοθεσία. Για το ECR, ο κύριος Βόντρα. Ευχαριστώ. Εγώ προέρχομαι από τη συντηρητική παράταξη η ομάδα μας έχει, κόμμα, έχει μέλη από την Πολωνία, Τσεχία, Ιταλία, χώρες με ενεργοβόρες βιομηχανίες. Και έχω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν, ως προς τη χαλιβουργία, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις. Αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, υψηλότερο κόστος παραγωγής άνθρακα από ό,τι σε τρίτες χώρες, και επίσης ε, μια χαμηλότερη επίδοση της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας, κάτι που απειλεί την επιβίωση της χαλιβουργίας στην Ευρώπη. Πρώτη ερώτηση. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χαλιβουργίας και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε πολυμερές επίπεδο. Μάλιστα υπάρχει μια παρατήρηση ε, στο παράρτημα του New Green Deal, ότι, ώστε μέχρι το 2030 να έχουμε διαδικασίες παραγωγής χάλιβα με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Πώς θα Μπορείτε να μας διευκρινίσετε πώς θα το υλοποιήσετε αυτό. Επίσης, χάλιβα χρειαζόμαστε και για να και για το στρατό, στρατιωτικό εξοπλισμό και για τα αυτοκίνητα. Ασχολείστε και έχετε στο χαρτοφυλάκιό σας και την άμυνα. Ε, σίγουρα εμπορικό πόλεμος ε, κίνα είπα, ίσως δημιουργήσει προβλήματα και εντάσει παγκοσμίω. Ένα λόγος παραπάνω λοιπόν να προσπίσουμε την ευρωπαϊκή χαλιβουργία. Για πολλούς από εμά επίσης είναι αδύνατο να υλοποιήσουμε αυτή την ενεργειακή μετάβαση χωρίς χρήση πυρηνικής ενέργειας. Εδώ όμως στην Εύη, έχουμε σαφώς ε, ε, αντιπροσωπείες που είναι κατά της πυρηνικής ενέργειας. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε μια πιο φιλοπεριβαλλοντική πυρηνική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε με κρατικές ενισχύσεις. Και μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας για τις κρατικές ενισχύσεις στην ατομική ενέργεια. Παρόμοια ρώτησαν άλλοι για τα χημικά. Έπρεπε εγώ να είχα μιλήσει για τα πυρηνικά, το ξέχασα πριν. Ο Μικ για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Επίτροπο για την παρουσίασή του. Έχω σοβαρές επιφυλάξεις ε, για το αν μπορούμε να υλοποιήσουμε την ε, δίκαιη μετάβαση με τις ελεύθερους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες. Εμείς έχουμε τεράστιους τυρφώνες στην Ιρλανδία που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Και η χρήση της τύρφης μέχρι το 2023 θα πρέπει να καταργηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θα πλήξει την Ιρλανδία. Η Ιρλανδική κυβέρνηση έχει προτείνει δύο σχέδια ε, για να α, αποζημιώσει όσους έχουν απολυθεί, έχουν χάσει τη δουλειά τους που, που είχαν από την συγκομιδή τύρφης για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Βέβαια, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα ευοδοθεί αυτό το σχέδιο λόγω των κανόνων ε, ε, δημόσιας, ε, δημοσίων συμβάσεων και του ανταγωνισμού που υφίστανται οι Ιρλανδικές επιχειρήσεις. Ίσως θα πρέπει να έχουμε καλύτερα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Βέβαια, δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο, κυρίως για πιο ηλικιωμένους εργαζομένους, που είναι δύσκολο άνθρωποι κάποιες ηλικίε να αναπτύξουν νέε δεξιότητε Και λόγω των κανόνων για τι δημόσιες προμήθειε, ακόμη και αν ε, να αναπτύξουμε νέε καλλιέργειε σε κάποιου εργαζόμενου. παρόλα αυτά, η επαγγελματική του σταδιοδρομία στο μέλλον θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Οπότε, πολλοί τέτοιοι εργαζόμενοι δεν θα έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία λόγω των ε, κανόνων που ισχύουν για τι κρατικέ ενισχύσει και τι δημόσιε προμήθειε. Αν θέλουμε δίκαιη μετάβαση, θα πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο κάποιους κλάδους, ε, κυρίως ε, σε χώρες όπως η Ιλλανδία, που θα επηρεαστούν ιδιαίτερα από τη δική μετάβαση. Και το Green Deal του Δεκεμβρίου είπε ότι θα αναθεωρηθούν ε, οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις μέχρι το 2021 για να ανταποκριθούν στους στόχους της Νέας Πράσινης Συμφωνίας. Εσείς κύριε Επίτροπε, πώς θα αναθεωρήσετε τους κανόνες αυτούς για τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες προμήθειες μπορείτε να καθησυχάσετε εμένα και τους Ιρλανδούς εργαζόμενους που φοβούνται θα χάσουν τη δουλειά τους και που εκπροσωπώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον Επίτροπο για 10 με 12 λεπτά για να απαντήσει στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων και θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συντονιστές για τις ερωτήσεις τους. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις του κυρίου Πίτερ Λίζε που αφορούσαν τις κρατικές ανισχύσεις και τις φιλοδοξίες για το περιβάλλον. Είπα ότι στην αναθεώρηση των κανόνων ανταγωνισμού θα ληφθούν υπόψη οι στόχοι μας για το περιβάλλον και το κλίμα. Και θα συζητήσω με την συνάδελφο Φερστάγκερ ώστε να εξετάσουμε τους κανόνες ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δεύτερη ερώτησή του ήταν πιο τεχνικής φύσεως. Μιλήσατε για χημικά προϊόντα που περιλαμβάνονται σε πλαστικές ύλες. Μιλήσατε κυρίως για το μόλιβδο. Αν κατάλαβα καλά. Σημαντικός αυτός ο στόχος, όντως. Πάντως, εμείς ζητήσαμε μείωση του μολύβδου στα πλαστικά εφαρμογή της οδηγίας REACH για να προστατεύσουμε την υγεία και το περιβάλλον. Και η σχετική εξαίρεση ήταν απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί ε, αυτή η παρακαταθήκη που είχαμε από το παρελθόν. Πάντως, τα πλαστικά που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε μόλιβδο ε, θα πρέπει να υποβληθούν σε ανακύκλωση. Και από τη μετάβαση στο 1 στα 2% 27 τόνοι μολύβδου μπορούσαν να εκλειθούν στο περιβάλλον. Είχαμε εκφράσει τις απόψεις μας ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μπαλάκι είναι τώρα στο δικό σας ε, γήπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Οπότε θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Στη συνέχεια, ερωτήσεις έθεσε η κυρία Γιούτελαντ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Έτσι δεν είναι. Μιλήσατε για την ηλεκτροδότηση και την ανάγκη να έχουμε ευρύτερη κάλυψη των υποδομών. Αυτό θα το συζητήσω στην Επιτροπή με τον κύριο Τίμερμανς, γιατί χρειάζεται και η δική του συμβολή. Είναι ένα κέριο ζήτημα αυτό. Και όταν προηγουμένως μίλησα για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, είπα ότι δεν μιλούμε πια για δισεκατομμύρια, αλλά για τρισεκατομμύρια δεδομένης της ε, διάρκειας του σχεδίου. Φυσικά θα έχουμε τεράστια, τεράστιες οικονομικές προκλήσεις, θα στηριχτούμε και σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τομέα αυτό, αν θέλουμε να υλοποιήσουμε όντως το στόχο της δίκαιης μετάβασης. Συμφωνώ με την ανάλυση σας και θα προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε όσο δυνατό περισσότερα μέσα και κονδύλια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς. Πάντως, συμφωνώ μαζί σας για την αλληλέδατα αυτά που επισημάνατε. Για την ανάγκη εναρμόνιση των κανόνων τώρα, φυσικά και στερνιζόμαστε αυτό το στόχο. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα του νομοθεσία REACH για τις χημικές ουσίες. Λαμβάνουμε υπόψη βέβαια τι ιδιαιτερότητε του κάθε κλάδου, αλλά απότερο στόχο μα είναι μια εναρμόνιση προ το συμφέρον τη αγοράς. Τρίτη ερώτηση. Το κύριο Τόρβαλτς. Άκουσα με μεγάλη προσοχή το σχολιά σας για το σχέδιο Φώσταν. Κρίμα που δεν πήγα και εγώ μετά από αυτά που μας περιγράψατε. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον το σχέδιο αυτό. Τώρα για τα open source. Καταπληκτικό το σχέδιο του open source. Πιστεύω ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και έμαθα από εσάς ότι παρόλο που βρίσκεται στις Βρυξέλλες αυτό το σχέδιο δεν έγινε καμία μνήα του. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι αν οι οργανωτές με καλέσουν του χρόνου θα πάω οπωσδήποτε. Σίγουρα θα μας ε, ενδιαφέρει στο μέλλον ιδιαίτερα αυτό το σχέδιο. Και μια και ε, υπάρχουν ε, δεσμοί με επιχειρήσεις που αναφέρεται, ένα λόγο παραπάνω. Θα το αναθέσω στο γραφείο μου να το φροντίσει. Η κατάσταση της οικονομικής ανάπτυξη και εγώ διαβάζω αυτό το συγγραφέα, είναι από τους αγαπημένους μου. Τώρα, τι προσπάθειες θα πρέπει να κάνουμε και τι εξελίξεις να επιδιώξουμε. Εδώ θα είχαμε δύο ερμηνείες. Καταρχήν μία από το πρίσμα της τεχνολογικής επανάστασης, γιατί μιλήσαμε για τα ψηφιακά θέματα, για την ψηφιοποίηση που αλλάζει και τη συμπεριφορά μας απέναντι στα διάφορα προϊόντα και θα χρειαστεί και αλλαγή των οικονομικών κανόνων και πολύ σημαντικοί οικονο... οικονομολόγοι, μερικοί έλαβαν και το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας, συνδυάζουν αυτή την οικονομική πραγματικότητα με την ε, νέα άειλη πραγματικότητα. Θα, θα πρέπει φυσικά αυτό να το λάβουμε υπόψη. Και επίσης να δούμε τι κονδύλια θα χρειαστούν. Και είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί όταν έχουμε ψηλά επίπεδα χρέους ίσως επηρεάσει το ηθικό, των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και ολόκληρα, ολόκληρους κλάδους. Και φυσικά υπάρχει το χρέος του παρελθόντος, που είναι αυτό που κληροδοτούμε στα παιδιά μας, αλλά υπάρχει το χρέος του μέλλοντος. Είναι τι πλανήτη θα αφήσουμε στις επερχόμενες γενιές. Και χωρίς ε, νέα πράσινη συμφωνία είναι σαν να λέμε στα παιδιά μας, όχι μόνο θα πληρώσετε τα σπασμένα του παρελθόντος, αλλά θα αναλάβετε και τα σπασμένα του μέλλοντος. Οπότε έχουμε μια ηθική ευθύνη, ηθικό καθήκον. Ε, και πραγματικά θα ξαναδιαβάσω το βιβλίο που αναφέρατε. Και νομίζω ότι ρόλος μας είναι και πέραν των οικονομικών μας υποχρεώσεων είναι να θεσπίσουμε κάποιες κανόνες για να λάβουμε υπόψη αυτό το χρέος του μέλλοντος και να το διευθετήσουμε τώρα για να μην το αφήσουμε κληροδότημα στις μελλοντικέ γενιές. Μετά, ε, ερωτήσατε η κυρία Μπενιέ. Ε, κατάλαβα αυτά που είπατε. Σε μερικά συμφωνώ, σε άλλα όχι. Συμφωνώ με αυτό που για την προκαθορισμένη παλαίωση. Αυτό είναι τμήμα της κυκλικής οικονομίας. Και συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας ε, και να δούμε τι θα περνάει από τα σύνορά μας. Εγώ ο ίδιος μίλησε για τον ε, ε, συνοριακό φόρο άνθρακα για να αποφύγουμε ακριβώς τέτοιες τρευλώσεις και επιζήμιες συνέπειες για τη βιομηχανία μας. Φυσικά μας ενδιαφέρει αυτό. Βέβαια, έχουμε σημαντικές σχέσεις με τους εταίρους μας και θα πρέπει και αυτές να τις λάβουμε υπόψη. Τώρα, αντίκτυπο στους πολίτες. Φυσικά θα πρέπει να βοηθήσουμε όλες τις ε, περιοχές και φυσικά να μην πληρώσουν την ύφη της μετάβασης οι πολίτες. Γι' αυτό ακριβώς φροντίσαμε το νέο πράσινο σύμφωνο να είναι τόσο φιλόδοξο. Και μετά μιλήσατε για το νεοφιλελεύθερο δόγμα. Έγιναν όμως κάποιες αλλαγές όπως θα διαπιστώσατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει κυρίαρχη όλο και περισσότερο σε κάποιους τομείς. Μιλήσαμε για κάποιες κέρδες τεχνολογίες, νευραλγικές, αλλά και για τους κρίσιμους πόρους ή τον, ε, τους ε, στρατηγικούς μας ανεφοδιασμούς, σπάνιες γέες για παράδειγμα ή τέτοιες σπάνιες πρώτες ύλες. Και μέχρι στιγμής, επειδή αντιλούσαμε τέτοιους πόρους ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αξιοποιήσαμε δεχομένω ή δεν διαρευνήσαμε τους δικούς μας. Ίσως στο μέλλον θα πρέπει να το κάνουμε. Και ε, για, για το 5G θέλουμε κανόνες, όπως και σε άλλους τομείς, που θα είναι εύληπτοι, ευανάγνωστοι, ώστε όσοι θέλουν να, να συνεισφέρουν να το κάνουν, αλλά με βάση τους δικούς μας κανόνες και όχι κανόνες που θα επιβάλλονται έξωθεν. Ο κύριος ε, Ζαντού. Είχατε μια ερώτηση καταρχάς. Τι ήταν η ερώτηση. Α, το πρότυπο γύρω 7. Οι αλλαγές των κανόνων για τα αυτοκίνητα ανεπαρκείς κανόνες, ε, πώς θα βοηθήσουμε την απομάκρυνση από τους ε, παραδοσιακούς κινητήρες ε, καύσεως. Κοιτάξτε, ο στόχος που μοιραζόμαστε είναι να έχουμε ένα όχημα μηδενικών εκπομπών. Εγώ το λέω ανοιχτά ως επίτροπος αυτός είναι ο στόχος μου. Τώρα, έχουμε θέσει μια φιλοδοξία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Θα πρέπει ε, αυτός ο στόχος ε, να, να τον συμμερίζονται οι περισσότεροι δυνατοί πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτά που αναφέρατε για τα αυτοκίνητα diesel, αλλά και τα βενζινοκίνητα νομίζω Δανία, Ισπανία, κάτω χώρες ε, και άλλες χώρες είχαν θέσει ένα στόχο, έναν ορίζοντα 2035-40 ίσως. Όλες αυτές είναι θαυμάσιες πρωτοβουλίες και σίγουρα θα τα προσέξουμε και θα τα συνοδεύσουμε αυτές τις διαδικασίες, τους στόχους, αυτές τις προσπάθειες των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να ισορροπήσουμε μεταξύ, αν θέλετε, των δύο αυτών κατευθύνσεων και θα χρειαστώ και τη βοήθειά σας. Γιατί όσο περισσότεροι συμμετέχουμε, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς που μας θυμίσετε και εσείς. Αλλά επαναλαμβάνω, ο επίσημος στόχος μας είναι τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Euh, euh, euh, Ο κύριος ε, Βόντρα για το χάλιβα. Στρατηγική ε, σημασίας ε, κλάδο, το θυμήσατε και εσείς, και για τα αυτοκίνητα αλλά και για την άμυνα. Είναι προφανές ότι εμείς θα προστατεύσουμε τη βιομηχανία αυτή στην Ευρώπη και όταν μιλούσαμε για την προσαρμογή ε, του άνθρακα στα σύνορα, μιλούσαμε πάνω απ' όλα για τα θέματα μεταλλουργίας. Αλλά δεν περιμέναμε δηλαδή, αυτό προσπαθώ να πω. Κοιτάξαμε να δούμε τι λύσεις μπορούμε να προσφέρουμε τι απαντήσεις μπορούμε να, μπορούμε να δώσουμε. Ε, τώρα θα πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνολογική καινοτομία και θα πρέπει να συνοδεύσουμε να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα πράγματα, την πρόσβαση στην αγορά, τις κρατικές ενισχύσεις, έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε εφόσον θα είναι απαραίτητο. Έχουμε εργαλεία, έχουμε τρόπους. Αυτό είχε πάντω ρητά αναφερθεί και συζητηθεί και στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Νομίζω ότι επίσης είχαμε ποια άλλη ερώτηση. Ο κύριος Βουάλλα. Είχα μια έτσι αφευγαλαία εντύπωση ότι είστε Ιρλανδός, δεν είναι. Δεν ήταν ερώτηση η δική μου, αλλά επειδή μιλήσατε για την τύρφη και τη συγκομιδή της, ε, πρέπει να πω ότι είναι ακριβώς αυτή μια περίπτωση, ένα παράδειγμα, όπου, όπου χρειάζεται να συνοδεύσουμε, να προστατεύσουμε αυτήν την μεταβατική διαδικασία, την προσπάθεια και να είναι δίκαιη. Αυτό είναι σημαντικό διότι ε, μας το θυμήσατε σε όλες τις διαστάσεις του, πρέπει να έχουμε κατά νου ε, και τους ανθρώπους εκείνους που θα απομακρυνθούν από τα επαγγέλματα αυτά, που θα ανακαταρτιστούν, πρέπει να γνωρίζουμε και να προσφέρουμε λύσεις και για αυτές τις περιπτώσεις εργαζομένων. Ε, χρειάζονται στηρίγματα, χρειάζεται υποστήριξη και κρατική υποστήριξη, από οποιαδήποτε δυνατότητα παρέμβαση μπορεί να έχει η Επιτροπή. Και θυμίζω ότι το Ταμείο ε, μπορεί να κινητοποιήσει μέχρι και 100 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι αμεληταία ποσά. Και αναφερόμαστε σε συγκεκριμένε περιπτώσεις όπως αυτή που αναφερθήκατε κι εσεί. Όλου δηλαδή εκείνους τους ανθρώπους που εργάστηκαν σε αυτόν τον κλάδο μια ολόκληρη ζωή. Είναι δύσκολο να προσφέρουμε επανακατάρτιση σε όλους αυτούς. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική βεβαίως. Πάντως, γι' αυτό προβλέψαμε ένα ειδικό κονδύλι, ένα ειδικό ταμείο, μπορεί να έχουμε και άλλα, για αυτό το μεγάλο έργο βοήθειας και υποστήριξης αυτών ακριβώς των μεταβατικών περιπτώσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Παρακαλώ να περιοριστείτε στο ένα λεπτό γιατί μας έχουν απομείνει 20 λεπτά με τον Επίτροπο. Οπότε για να μπορέσει να απαντήσει ε, θα πρέπει να το αφήσουμε και χρόνο. Ξεκινάμε με το ΕΛΚ και την Εστέρ Ντελάνγκε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, στην εισαγωγή σας μιλήσετε για παγκόσμιο ηγετικό ρόλο και πράσινη τεχνολογία, πράσινους πρωταθλητές θα λέγαμε. Βεβαίως για το ΕΛΚ αυτό δεν σημαίνει εταιρείε που καθορίζουν οι πολιτικοί, αλλά αναδεικνύονται από τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός ο οποίος πρέπει να είναι δίκαιος όμως. Μιλήσατε πολύ για κρατικές ενισχύσεις ε, για εμάς δεν είναι αυτή η πλήρης εικόνα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από την Ολλανδία όπου κάνουμε δημόσιες προμήθειες για πράσινες ε, μαζικές μεταφορές, δηλαδή ηλεκτρικά λεωφορεία όπως ακριβώς θέλουμε και τελικά προέκυψε ότι η εταιρεία η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό θα κατασκευάσει τα περισσότερα λεωφορεία στην Κίνα όπου εμείς όμως δεν έχουμε πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες της Κίνας, οι περισσότερες εταιρείες εκεί έχουν κρατικές ενισχύσεις κτλ. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξής. Σας λέω αυτό το παράδειγμα γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι εάν το πράσινο deal σημαίνει ότι θα αγοράζουμε όλα αυτά τα πράσινα αγαθά και υπηρεσίες από την Κίνα, δεν θα λειτουργήσει. Οπότε δεν πρέπει να συζητάμε μόνο τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά και τις δημόσιες προμήθειες θα είμαστε σε θέση να αποκλείουμε από τις δημόσιες προμήθειες εταιρείε από χώρε που δεν μας επιτρέπουν πρόσβαση στην αγορά τους. Πρέπει να έχουμε και την εργαλειοθήκη κατά του dumping. Θυμηθείτε τι συνέβη με τα ηλιακά πάνελ από την Κίνα. Ε, η τεχνολογία που αναπτύσσεται εδώ και μετά βγαίνει εκτό αγορά. Είστε διατεθειμένο ω επίτροπο, παραδείγματο χάρη, να κάνετε συγκεκριμένε νομοθετικέ προτάσει για τι δημόσιε προμήθειε. Γιατί ε, έχει αργήσει, θα έλεγα. Ευχαριστώ κυρία Μόζελ για τους σοσιαλδημοκράτες. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Θα ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα πως χαίρομαι που ακούτε ότι είναι καλή ιδέα το ότι η Ολλανδία και η Δανία θέλουν να παγορέψουν τα οχήματα ντίζελ από το 2030, τα γιοταχή. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Μίληστε για μια κατάσταση ανταγωνισμού, ο οποίος θα είναι δίκαιος για τις ευρωπαϊκές ε, εταιρείε. Το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για την ανταγωνιστικότητα παγκοσμίω ε, είναι να είμαστε φιλόδοξοι και να έχουμε υψηλέ απαιτήσει. Λοιπόν, εδώ. Μπορείτε να ανεβάσετε τις προδιαγραφές του Euro 7. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και να προχωρήσουμε έτσι ώστε να προχωρήσουν κάποιοι για να έχουμε την δυνατότητα να επιβιώσουμε στον ανταγωνισμό. Σας ευχαριστώ για το ρηνιού. Βερονίκ Τριγέ Λενοάχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα σας μιλήσω γαλλικά. Και θα σας μιλήσω για κάτι που εντάσσεται στον οδικό σας χάρτη, την τεχνητή νοημοσύνη και την εφαρμογές της στον τομέα της υγείας η συνδυασμένη εφαρμογή ε, των μαζικών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στο ανθρώπινο γονιδίωμα επέτρεψε σημαντική πρόοδο στην θεραπεία για καρκίνο στην ιατρική και στην πρόληψη μεγάλου αριθμού νόσων. Βέβαια θα πρέπει να αποφύγουμε πιθανή εκτροπή αυτής της κατάστασης γιατί όχι μόνο θα δημιουργήσουμε διακρίσεις στην απασχόληση και στις ασφάλειες, αλλά έτσι φαίνεται ότι μπορούν να προβλεφθούν και νέα, νέα είδη συμπεριφορά. Κυρίω το κοινωνικο-οικονομικό, οικονομικη θέση, ο χρόνος στο σχολείο ή σεξουαλικός προσανατολισμός. Αυτά πραγματικά θα ήταν ε, στρεβλές εφαρμογές που θα δημιουργούσαν σε μια τεχνολογική ε, ευγονία πώς θα βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των κινδύνων που ενέχουν οι νέε τεχνολογίες και των ευκαιριών που είναι αναφυσβήτητε ε, από τη χρήση του ιδιαίτερα στον τομέα τη υγεία. Ευχαριστώ. Για το ΕΛΚ, η κυρία Τότς. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε. Σα ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυναμική βιομηχανία η οποία παίζει έναν ε, ρόλο κλειδί στην οικονομία μας. δουλειά σας είναι να διασφαλίσετε πως όλα τα κομμάτια της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα συνεισφέρουν εξίσου σε μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Προσεχώς ε, θα παρουσιάσετε μια ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για να δούμε το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας ε, νέες δουλειές και επενδύοντας στην πράσινη τεχνολογία. Άρα η ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση και ο μόνος τρόπος ε, να διασφαλίσουμε ότι η πράσινη μετάβαση ε, δεν θα οδηγήσει σε διαρροή άνθρακα και απώλειες θέσεων εργασίας. Οπότε πρέπει να συνδέσουμε το πράσινο deal με μια στιβαρή βιομηχανική πολιτική που θα κινητοποιήσει τις απαραίτητες επενδύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω πώς θα δει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής η βιομηχανική πολιτική ενισχύοντα την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Ευχαριστώ για το ID Casting Κρίζα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επιτρόπε, αναφερθήκατε στην μετανάστευση υπό την οικονομική σκοπιά. Αλλά μια τέτοια σκοπιά δεν λαμβάνει υπόψη της τις περιβαλλοντικές συνέπειες του φαινομένου αυτού. Περισσότερη κατανάλωση σημαίνει περισσότερη παραγωγή και επομένως περισσότερη ρήπανση. Χρειαζόμαστε λοιπόν υποδομές, ε, περισσότερες κατοικίες, ε, περισσότερη χρησιμοποίηση σκυροθέματος με όλες τις επιπτώσεις που ενέχει καθότι έχουν, και η Συμφωνία των Παρισίων έχει δείξει τα όρια της, είναι ε, τα δύο ε, αυτά στοιχεία ε, δεν μπορούν να συμφιλιωθούν αν θέλετε σε πλαίσιο οικολογικής στόχευσης και επομένως επίτροπε πώς μπορούμε να προωθήσουμε και τους δημογραφικούς μας αναπτυξιακούς στόχους αφενός και αφετέρου να προστατεύσουμε για το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Ένα θέμα που ίσως ε, ακόμα δεν έχει τεθεί στην Επιτροπή μας. S&D, ε, κυρία Μορέτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πολύ χαίρομαι και φαντάζομαι όλοι μας χαιρόμαστε που ακούμε να βεβαιώνεται ότι η Πράσινη Συμφωνία θα είναι η μεγαλύτερη φιλοδοξία για αυτήν εδώ την Επιτροπή και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς θέσαμε έναν στόχο πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να επιτύχουμε, να υλοποιήσουμε αυτό το νέο ευρωπαϊκό όνειρο. Να γίνουμε δηλαδή αυτό που εσείς ήδη μας ονομάσατε, μας περιγράψατε ως ηγετική δύναμη πράσινη στον κόσμο, αυτό θα αφορά μια ολόκληρη γενναία. Και θα είναι μια τεράστια προσπάθεια. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την ηγετική θέση και στις πράσινες τεχνολογίες, και εδώ μιλάτε για κυριαρχία πράσινες θα χρειαστούμε έρευνα και καινοτομία. Εσείς πώς σκοπεύετε να προωθήσετε και να υποστηρίξετε την ερευνητική προσπάθεια και την κατάρτιση. Η βιωσιμότητα πέραν των όσων ήδη ακούσουμε πρέπει να προωθήσουμε προγράμματα εκπαιδευτικά και ψηφιακά προς τους πολίτες και τους καταναλωτές και θα πρέπει να συνοδεύονται οι καταναλωτές, να, να πλαισιώνονται στις επιλογές που κάνουν ε, και θα, δεν θα πρέπει να μιλούμε μόνο για τα καταναλωτικά αγαθά αλλά και τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πολίτες. Θα ήθελα και γι' αυτό να μας πείτε κάτι λοιπόν σχετικά με τη φιλοδοξία της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Χαουτ για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Εδώ είμαι στα δεξιά σας να... Ε, στα αριστερά όπως κοιτάτε εσείς ε, ευτυχώς, εντάξει. Στα, στα τέρμα αριστερά, εντάξει. Ε, κοιτάξτε, αυτό δεν, δεν το έκανα εγώ, έτσι ήταν, έτσι. Λοιπόν, το σημαντικό είναι λέει το Κοινοβούλιο ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μειώσει το συνολικό της αποτύπωμα στο περιβάλλον και στους ε, πόρους. Ε, πώς θα το ενσωματώσετε αυτό τον στόχο μείωσης του συνολικού αποτυπώματος στο συνολικό σας ε, βιομηχανικό πρόγραμμα και τέλος θέλουμε να δούμε έναν κύκλο ε, των μη τοξικών υλικών και μέχρι τώρα η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης δεν κάνει κάτι για τα μη τοξικά υλικά. Ε, νομίζω είναι μάλιστα αντικείμενο των περισσότερων υποθέσεων στο δικαστήριο κατά τις Κομισιόν μόλιβδος, ενδοκρινικοί διαταράκτες λοιπά. Πώς θα αναπτύξετε λοιπόν έναν ε, κύκλο μη τοξικών υλικών και να μην παρατείνετε η χρήση των τοξικών υλικών. Σας ευχαριστώ για το έλκη κυρία Σπυράκη. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Είμαστε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά ασχολούμαστε και με θέματα δημόσιας υγείας. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να εστιαστώ στην βιομηχανική σας πολιτική και να σας ρωτήσω. Προσπαθείτε να αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε να, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα έλλειψης φαρμάκων, έλλειψης σκευασμάτων, ώστε να έχουμε παρκή φάρμακα και σκευάσματα για όλους τους ασθενείς. Αυτό αφορά άμεσα στις κρατικές ενισχύσεις στο φαρμακευτικό κλάδο στην Ευρώπη. Ε, φαντάζομαι ότι θα γνωρίζετε τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε στην εξωτερική ανάθεση προ τρίτε χώρες οι οποίες έχουν και αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που συχνά αναφέρουμε. Σα ευχαριστώ. Για το ECR, ο κύριος Φόντρα και πάλι, εκτός αν όχι, ε, ωραία. S&D. Αν θέλετε, παρακαλώ, παρακαλώ, μπορείτε. Μπορείτε δύο φορές να τοποθετηθείτε. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ δεν έλαβα απάντηση με το δεύτερο ζήτημα που έθεσα και με την άδειά σα το ξαναθέτω. Είναι αδύνατον για πολλούς από μας να περάσουμε αυτή την ενεργειακή μετάβαση χωρίς, την πυρηνική ενέργεια. Καλώς όλα αυτά που λέει ο Πίτερ και άλλοι για τα χημικά, αλλά το θέμα των κρατικών ενισχύσεων στην πυρηνική ενέργεια, πώς το απαντάτε, Επιτρόπε. Μάλιστα. Τίμο Βόλκεν, S&D. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, Όπω τον προλαλήσαντα υπάρχει η ατομική ενέργεια και λειτουργεί μια χαρά στην ε, Γερμανία. Έχω κάποιες ερωτήσεις, ε, κύριε Επιτροπέ, χαίρομαι που ήρθατε. Θα εξηλεκτριστούν πάρα πολύ κλάδοι. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε για όλους. Για όλους θα χρειαστούμε υδρογόνο και πράσινο υδρογόνο. Ακούσαμε πάρα πολλά σήμερα, αλλά όχι συγκεκριμένα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας θέσω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Έχει η Κομισιόν συγκεκριμένους αριθμούς για την ζήτηση πράσινου υδρογόνου για την ευρωπαϊκή οικονομία, ειδικά για την βιομηχανία για τα έτη 2030, 40 και 50. Και θα ήθελα να γνωρίζω ποια μέτρα θεωρείται αυτή τη στιγμή απαραίτητα για να είναι ανταγωνιστικό το πράσινο υδρογόνο και να περάσουμε από το φυσικό αέριο στο πράσινο υδρογόνο χωρίς προβλήματα και να δούμε παραδείγματο χάρη τι επενδύσει σε αγωγού αερίου έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το υδρογόνο για να μην ε, χρησιμοποιούμε συνεχώς την ενδιάμεση τελικά τεχνολογία του φυσικού αερίου. Σας ευχαριστώ για το Renew. Ευχαριστώ Πρόεδρε. για την ε, χρησιμοποίηση των τεχνολογιών νέας γενιάς όπως την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει η Ευρώπη να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις και θα πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς από μια βιομηχανική στρατηγική και να αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και επομένως χρειαζόμαστε μια, έναν ενιαίο χώρο, ε, ένα ενιαίο πλαίσιο για την διαλειτουργικότητα των δεδομένων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη δημόσια υγεία, την ενέργεια. Αυτός ο χώρος θα πρέπει να είναι εκτός για τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές, όπως και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για να μπορούν να κοινοτομήσουν. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε, αγαπητέ Επίτροπε, ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για μια πλήρως λειτουργική αγορά για τα δεδομένα και για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και ανωνυμοποίηση των δεδομένων, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογική κοινοτομία που πολύ χρειαζόμαστε και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Πώς θα προετοιμάσουμε λοιπόν την ηγετική θέση της Ευρώπης ε, στην ε, ε, ανάπτυξη που μας χρειάζεται για να πετύχουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και τα ηθικά πρότυπα και τη συνοδεία που χρειάζεται να συνοδεύσει την προσπάθεια αυτή. Ελκ, ε, Στάνισναφς Μπορσάκ, λέει ο Πρόεδρος, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση για την ε, ενιαία εσωτερική αγορά και τη νέα πράσινη συμφωνία. Θα πρέπει να αναλύσουμε όλες τις συνέπειες που θα έχει ενδεχομένω αυτή η συμφωνία στην εσωτερική αγορά και κυρίως στις επιχειρήσεις μας, αλλά και στους καταναλωτές. Όπως είπατε, θα υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις που με προβληματίζουν κάπως. Και θα ήθελα να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Την διτή ποιότητα των προϊόντων. Ε, αφορά τους καταναλωτές, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας τροφίμων. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία εγκύψαμε σε αυτό το θέμα. Τα, προϊόντα, τα ίδια προϊόντα, ανάλογα με το σε ποια χώρα ε, διατίθενται σε εμπορία, έχουν διαφορετική ποιότητα. Έτσι δημιουργούμε δύο κατηγορίες αγορών, τη δυτική αγορά και την ανατολική αγορά και στη δυτική αγορά τα προϊόντα έχουν καλύτερη ποιότητα. Είναι απαράδεκτη αυτή η διπλή ποιότητα προϊόντων. Είστε αρμόδιος και για την εσωτερική αγορά. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτά τα διπλά μέτρα και σταθμά, αυτή τη διαφορετική ποιότητα που έχουν τα ίδια τρόφιμα ανάλογα με το σε ποια χώρα διατίθενται. Αυτό είναι άδικο για τους καταναλωτές και τους φέρνει σε δυσμενή θέση, κυρίως σε τους καταναλωτές της Ανατολικής Ευρώπης που αγοράζουν προϊόντα χειρότερης ποιότητας. Αυτό το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες και ήταν σημαντικό στοιχείο και της προεκλογικής συζήτησης στη Ζεχή αλλά και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Κόκαλης, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δεν είμαι βέβαιος ότι η φάση της οικονομικής ανάπτυξης του Ρώστο μας ενδιαφέρει τόσο σε αυτήν την εποχή της ραγδαίας εξέλιξης. Τη στιγμή που ε, το, το ρολόι της έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ε, είναι αντιφατικό μερικές φορές με την ανάγκη της μετάβασης. Ε, πώς θα αποφύγουμε λοιπόν να εγκλωβιστούμε ε, σε επενδύσεις ε, σε, ορυκτά, σε ορυκτό αέριο όπως είναι το φυσικό αέριο. Και ποιες είναι οι οικονομικές, κατά, κατά τη γνώμη σας, ευκαιρίες που δημιουργούνται από αυτή την ε, προσαρμογή στη νέα κατάσταση. Ευχαριστώ. Επισήμως να απομείνει δύο λεπτά από το χώρο που έχουμε προβλέψει. Άντε να τα κάνουμε 5-7 το πολύ για να προλάβει ο Επίτροπος να απαντήσει συνοπτικά όμως ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων και αρκετά πλούσια. Αν δεν προλάβω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις τώρα, θα σας στείλω γραπτός ε, απαντήσεις διμερώς αυτά που παρέλειψα. Σίγουρα οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι φάμιλες των φιλοδοξιών μας. Μιλήσαμε για τη δίκαιη μετάβαση σήμερα αλλά και με τους συναδέλφους, τον κύριο Τζεντιλόνη, ε, εξετάζουμε μηχανισμούς για πιο φιλόδοξες επενδύσεις, χρησιμοποιώντας και πιο μακροπρόθεσμα ομόλογα, αξιοποιώντας τα ε, εξαιρετικά επιτόκια που έχουμε σήμερα, που μερικές φορές είναι έως και αρνητικά. Έτσι θα δώσουμε μια καλύτερη όθηση και θα παρακολουθήσουμε και θα στηρίξουμε καλύτερα αυτή τη μετάβαση που είναι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο και θα απαιτήσει κινητοποίηση τεράστιων κονδύλιων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όλους τους ενδιαφερομένους. Και έχω επίγνωση αυτών των προκλήσεων και φυσικά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα για να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας. Θα ήθελα να καθησυχάσω την κυρία Τότ ότι σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαχωρίζει τους πολίτες της Ανατολικής ε, και Δυτικής Ευρώπης. Και το θέμα της διπλής ποιότητας των τροφίμων ε, είναι απαράδεκτο και θα φροντίσω στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μου να το αντιμετωπίσω. Επίσης για την πυρηνική ενέργεια που ακούστηκε τουλάχιστον δύο φορές. Ο κύριος που έθεσε την ερώτηση δυστυχώς δεν φοράει τα ακουστικά του και φοβάμαι ότι δεν θα με ακούσει ούτε τώρα και θα χρειαστεί να το πω και τρίτη φορά. Μιλάω για τα πυρηνικά, για την ατομική ενέργεια. Ευτυχώς που σας θυμήθηκα. Θυμήθηκα ποιος είχε υποβάλει την ερώτηση για τα πυρηνικά. Πολύ σημαντικό το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, πολύ σημαντική πηγή ενέργειας η πυρηνική για πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, θεωρείται μια μεταβατική ενέργεια η πυρηνική για την υλοποίηση του στόχου μας. Και σήμερα είναι εθνική αρμοδιότητα το θέμα αυτό του ενεργειακού μείγματος και όχι ευρωπαϊκή. Πάντως, η πυρηνική ενέργεια είναι ένα από τα στοιχεία του ενεργειακού μείγματος, αλλά η απότερη φιλόδοξή μας είναι να έχουμε μια οικονομία ε, καθαρή, καθαρής ενέργειας, χωρίς διοξίδιο του άνθρακα. Αλλά ως μεταβατική ενέργεια χρησιμοποιούμε και στην πυρηνική στο μείγμα. Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τα μαζικά δεδομένα, όντως ε, είναι σημαντική αυτή η τομής και αν με ξανακαλέσετε πολύ ευχαρίστως να επανέλθω για να σας παρουσιάσω τη λευκή βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα. Και η πρόεδρος μου ζήτησε να υιοθετήσουμε μια σφαιρική προσέγγιση για τη στρατηγική των δεδομένων, με τη ροή των δεδομένων, ώστε να έχουμε πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό δεδομένων και δημοσίων δεδομένων, αλλά όχι μόνο. Οπότε, σίγουρα είναι σημαντικό αυτό το θέμα και ήδη έχει ξεκινήσει η επεξεργασία του. Πάντως, ε, πολύ ευχαρίστω να έρθω μια άλλη στιγμή για να σα αναλύσω πιο διεξοδικά αυτά τα θέματα. Και οι ερωτήσει που μας θέσετε μας, βρίσκονται, μας βρίσκουν σύμφωνο και στα θέματα καινοτομία, ικανότητας έρευνας, πρόοδου και σε θέματα της χρήσης των δεδομένων που σε μεγάλο βαθμό θα παράγονται στην Ευρώπη. Και ο αλγόριθμος, οι αλγόριθμοι ελπίζω να ε, παράγονται επίση στην Ευρώπη και να χρησιμοποιούνται εδώ. Σε ό,τι αφορά το υδρογόνο, το πράσινο υδρογόνο, δεν έχω αριθμητικά στοιχεία συγκεκριμένα για να απαντήσω, γιατί αναφέρατε κάποια στοιχεία, αλλά θα εξετάσω αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω. Πάντω θέλουμε κάποια κοινά στοιχεία ευρωπαϊκού, ε, σχέδια ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και για το υδρογόνο. Και εγώ προσωπικά πιστεύω στο υδρογόνο και πιστεύω ότι θα έχει στρατηγική σημασία και θα μας επιτρέψει να λύσουμε πολλά προβλήματα των μεταφορών, της, της κινητικότητας και ούτω καθεξής. Τώρα για τα μη τοξικά στοιχεία. Και Εδώ έχουμε ένα πριν και ένα μετά. Θα έχουμε σαφείς κανόνες. Θα θεσπίσουμε σαφείς κανόνες. Και το έχω ήδη συζητήσει με τη Γενική Διεύθυνση Grow. Ήδη ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Κυρία Μωρέτη. ρώτησε για την έρευνα. Έχετε δίκιο. Θέλουμε να έχουμε τεράστιες ερευνητικές προσπάθειες και μεγάλη κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και χρειαζόμαστε φυσικά τα απαραίτητα κονδύλια και στην έρευνα. Και θα μας βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να παραμείνουν άθικτα τα κονδύλια για την έρευνα και το ορίζοντας 2020 και όλα τα συναφή προγράμματα έχουν συγκεκριμένα κεφάλαια ε, για το Green Deal και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην περικοπούν τα κονδύλια της έρευνας για να ανταποκριθούμε στις θεμητές ανάγκες που έχει η Ευρώπη σε θέματα έρευνας. Επίσης, ε, κάποιος από το ΕΛΚ, κάποια από το ΕΛΚ ρώτησε για τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία στις κάτω χώρες. Δεν το ήξερα ότι αγοράστηκα στην Κίνα και μάλιστα με πρότυπα που δεν ήταν παρεφερή με τα δικά μας και αυτό έγινε για να τηρηθεί ο διαγωνισμός. Πάντως θα προσπαθήσω να βρω λύσεις και μέσα, μηχανισμούς, ε, όπως η άμυνα, η εμπορική όταν υπάρχουν πιθανότητες του ανταγωνισμού. Θα δω τι μέσα έχουμε στο προστάσιό μας και πόσα μπορούμε να επικαλεστούμε και να εργοποιήσουμε. Τώρα, η αμοιβαιότητα στις δημόσιες προμήθειες. Το θέμα αυτό έχει κολλήσει στο Συμβούλιο από ό,τι ξέρω. Θα προσπαθήσω να το προωθήσω πάντως. Μέχρι στιγμής όμως υπάρχει αδιέξοδο στο Συμβούλιο για την αμοιβαιότητα στις δημόσιες προμήθειες. Πάντως, στα πλαίσια των κανόνων του ΠΟΕ, ε, χαίρομαι που μου το επισημάνατε, θα το διερευνήσω και θα το συζητήσω με τον ε, συνάδελφο Φιλ Χόγκαν. Νομίζω ότι απάντησα στους περισσότερους. Συγγνώμη, δεν τα κατάφερα να απαντήσω σε όλους. Κάποιος αναφέρθηκε στη μετανάστευση. Θέλουμε ικανότητες, θα τις δημιουργήσουμε όλο και περισσότερος για να υλοποιήσουμε το στόχο μας και θα αναπτύσσουμε τέτοιες ικανότητες και εσωτερικά και εξωτερικά. 450 εκατομμύρια είναι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και η φιλόδοξή μας για οικονομική ανάπτυξη είναι πάνω από 2% για να εξασφαλίσουμε και την κοινωνική μας πρόοδο. Και οι δημογραφικές προβλέψεις για το 2050 μας δείχνουν αμετάβλητο πληθυσμό μέχρι τότε, στα 350 εκατομμύρια δηλαδή, οπότε θα πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να υλοποιήσουμε και το στόχο του μηδενικού άνθρακα μέχρι το 2050. Όλα αυτά θα χρειαστούν για να προστατεύσουμε και τον πλανήτη μας που το 2050 θα έχει πια 9 δισεκατομμύρια από 7 δισεκατομμύρια κατοίκους που έχει σήμερα. Αυτά και θα σας στείλω γραπτό στις απαντήσεις που δεν κατάφερα να καλύψω γιατί δεν είχα χρόνο. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Euh, Ας κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα για να επανέλθουμε στο άλλο καυτό ζήτημα με το ECDC. Να επανέλθουμε, συνάδελφοι, αν θέλετε. Και προτού πάω στο θέμα του ECDC και να καλωσορίσω την εκτελεστική διευθύντρια ήδη, να κάνω μία-δύο ανακοινώσει για τη διάταξη, η πιο σημαντική των οποίων είναι ότι μετά το Brexit και την αποχώρηση των ε, Βρετανών μας συναδέλφων, αριθμητικά αλλάξαμε. Ε, αποφασίστηκε στην Ολομέλεια ότι η ΕΝΒΗ πλέον αποτελείται από 81 μέλη, αντί για 76 που ήταν μέχρι πριν. Είμαστε Έχουμε την αριθμητική σύνθεση, αλλά δεν έχουμε και τα ονόματα της νέας σύνθεσης, που θα εγκριθούν επισήμω στο Στρασβούργο την ερχόμενη εβδομάδα. Κάποιες πολιτικές ομάδες ζήτησαν να αναβληθούν αυτές τις ψηφοφορίες που ήταν να γίνουν σήμερα και συμφωνήσαμε να αναβάλουμε και να ψηφίσουμε επί του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου της νομοδότησης, της ε, έκθεσης, όταν θα έχουμε την πλήρη σύνθεση, τη νέα δηλαδή σύνθεση της Επιτροπής. Και θα έχουν εγκριθεί τα νέα μέλη στο Στρασβούργο. Αυτή είναι η βασική ανακοίνωση που είχα να σας κάνω. Και η κυρία Λενουάχ μου ζήτησε να αναφερθώ και στους επισκέπτες μας ε, από την Γαλλία. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ ή αν μας εγκατέλειψαν. Τέλο πάντων, η πρόθεσή μου ήταν να του καλωσορίσω θερμά. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στην δεύτερη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε σήμερα με το ε, Ευρωπαϊκό Κέντρο πρόληψη και Ελέγχου Νόσων. Η ετήσια συνάντησή μας είναι αυτή, αλλά βεβαίως έρχεται σε πολύ κέριο χρονικό σημείο με τον ιό κορώνα και θα ήθελα η Διευθύντρια να εστιαστεί κυρίως, όχι αποκλειστικά, στον κορώνα, να έχουμε τη δική σας δηλαδή αξιολόγηση του επίπεδου κινδύνου ή του τρόπου αντιμετώπισης εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς και επίσης αν θα μπορούσατε και στα πλαίσια της παρουσίασής σας να αναφερθείτε και σε άλλα ζητήματα, γιατί βέβαια το κέντρο πρόληψης δεν είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στον κορώνα. Έτσι. Λοιπόν, έχετε το λόγο για 10 με 15 λεπτά, κυρία Διευθύντρια, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με προσκαλέσατε σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων ε, με την Επιτροπή σας και ιδιαίτερος ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κοτσίνσκα που είναι η νέα Ευρωβουλευτής επιφορτισμένη με την επαφή μαζί μας και τους δύο εκπροσώπους ε, του Κοινοβουλίου, το Διοικητικό μας Συμβουλίο, την ε, Σοφία Κούκοβιτς και την ε, Μαριλένα Κουπά. Η ε, αυτή ακρόαση θα εστιαστεί σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα όμως να ευστήσω την προσοχή σας στο ότι παρά το ότι εστιάζουμε στον κορονοϊό, οι άλλοι ιοί και τα βακτηρίδια που απειλούν την ανθρώπινη υγεία στην Ευρώπη δεν κοιμούνται. Και σας διαβεβαιώ ότι συνεχίζουμε να τους παρακολουθούμε, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι τον περασμένο μήνα Δημοσιεύσαμε τέσσερις ε, αξιολογήσεις ε, κινδύνου για τον κορονοϊό και τρεις ε, άλλες. Δύο από αυτές ασχολούνται με παθογόνους παράγοντες που αντιστέκονται στα φάρμακα. Ένα μήνυμα δηλαδή για την άλλη απειλή την οποία θα σας παρουσιάσω σήμερα. Να προσπαθούν εδώ με τις διαφάνειες. Ακόμα. Λοιπόν, να δούμε λίγο το ιστορικό και το έτος 2003 τότε συζητούσαμε τον ιό SARS, επίσης κορονοϊό, που ήταν η αφορμή να ιδρυθεί το κέντρο μας. Σήμερα, μετά από 15 χρόνια, το κέντρο μας είναι μια υπηρεσία με προσωπικό 280 ατόμων από 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν ετήσιο προϋπολογισμό 60,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και βεβαίως ε, τώρα θα έρθω στον ε, κορονοϊό. Οι κορονοϊοί ταυτοποιήθηκαν ε, πριν από πολλά χρόνια στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και πως βάλουν ανθρώπους και κάποια ζώα. από το 2003 υπήρχαν ε, για τους, υπήρχαν κορονοϊοί που προσέβαλαν τους ανθρώπους, ο ΣΑΡΣ και ο ΜΕΡΣ. Ταυτοποιήθηκε δε ο νέος κορονοϊός ε, στα τέλη του 2019. Πρόκειται για ένα νέο στέλεχος, το οποίο δεν είχε ταυτοποιηθεί μέχρι τότε σε ανθρώπους. Ε, και βεβαίως κάτι τέτοιο είναι κάτι το οποίο πάντα είναι ενισχυτικό, ειδικά όταν δεν γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του ιού, το πώς ε, διαδίδεται και τι χαρακτηριστικά έχει η αρρωστία και πώς αντιμετωπίζεται. Εντάξει, έχει ανέβει ή όχι. Βλέπετε λοιπόν ε, τις ενδείξεις στο κέντρο επιχειρήσεων ε, ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σε επίπεδο συναγερμού 2. Το υψηλότερο επίπεδο δηλαδή που έχουμε ε, δουλεύουμε σε δύο βάρδιες το 24ωρο. Μπορούμε δηλαδή να δουλέψουμε και 24 ε, ώρες το 24ωρο. Τώρα πραγματικά είναι κρίμα που δεν έχω τη διαφάνεια γιατί θα ήθελα να σας δείξω έναν χάρτη. I don't think this was this. Okay, uh, maybe I can show you later. I um, uh, just wanted to uh, update you as of... Να σα ενημερώσω λοιπόν για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα το πρωί. Έχουμε 17.383 ε, περιπτώσει κρούσματα δηλαδή και 362 θανάτους. Η πλειοψηφία βρίσκεται στην Κίνα και όλοι οι θάνατοι στην Ασία, 361 στην Κίνα και ένας στις Φιλιππίνες. Στην Ευρώπη έχουμε 25 κρούσματα, 21 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 2 στη Ρωσία. Θα σας τα πω τα υπόλοιπα μετά. Υπάρχουμε, λοιπόν, μια, υπάρχει μια ιστοσελίδα που ενημερώνουμε καθημερινά ε, τις πληροφορίες ε, και φροντίζουμε έτσι να είναι ενημερωμένο το κοινό, όχι μόνο οι επαγγελματίες. Η αξιολόγηση κινδύνου χρησιμοποιείται από τα ΜΜΕ και τον τύπο και έχουμε πολλές επαφές ε, με τα ΜΜΕ. Η τρέχουσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 21 κρούσματα είναι πως ε, ο στόχος είναι να περιοριστούν τα κρούσματα αυτά και να μην υπάρξει περαιτέρω διάδοση. Οι συνάδελφοι εκεί το κάνουν αυτό μέσω της έγκαιρης διάγνωσης των κρουσμάτων, της απομπόνωσης ταυτοποίησης ε, όλων των επαφών που έχουν και βεβαίως ε, ενημέρωσης. Αυτό έχει γίνει. Από τα 21 κρούσματα αυτά έχουμε 8 ε, όπως είπα στην Γερμανία, ένα στη Γαλλία. Όλες οι άλλες, όλα τα άλλα κρούσματα είναι εισαγόμενα τρόπον την Οπότε η κατάσταση στην Ευρώπη είναι υποέλεγχο θα έλεγα. Αυτό θα το δούμε μετά. Ο στόχος λοιπόν είναι να βοηθήσουμε τις χώρες ε, να μην διαδοθεί περαιτέρω η αρρώστια. Και ακριβώς αυτό το στόχο έχει το οτιδήποτε παράγουμε ως υλικό. Πέρα λοιπόν από την αξιολόγηση κινδύνου, η τελευταία μάλιστα έγινε 20, 21 Ιανουαρίου. Συμφωνήσαμε στον ορισμό των κρουσμάτων σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ε, για το πώς θα βρεθούν οι επαφές και βεβαίως ε, μια εναρμονισμένη αντίδραση για το που θα πρέπει να καταυθύνονται οι ύποπτες περιπτώσεις για τεστ, πώς θα ειδοποιούνται οι οι επαφές και το τελευταίο έγγραφο το συντάξαμε το Σαββατοκύριακο και αφορούσε μέτρα πρόληψης ε, της διάδοσης ε, σε εγκαταστάσεις υγείας. Και μία από τις ε, δραστηριότητές μας για να δούμε ακριβώς ε, ποια είναι η ετοιμότητα των χωρών. Έχουμε κάνει μία μελέτη των εργαστηρίων για να δούμε αν οι χώρες είναι σε θέση να ανοιχνεύσουν τον ιό, που είναι βεβαίως η αφετηρία. Δεν έχω δει τα αποτελέσματα αλλά όπως ξέρουμε οι χώρες ε, μπορούν να ανοιχνεύσουν και υπάρχουν εργαστηριά σε πέντε κράτη-μέλη που έχουν την δυνατότητα να ε, ελέγξουν και τα δείγματα άλλων χωρών και θέλουν κιόλας. Επίσης ε, έχουμε αναπτύξει κάποια υποδείγματα, φυλάδια για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και για τους ταξιδιώτες. Ε, περιέχουν ένα κομμάτι για ταξίδια προς την Κίνα και από την Κίνα. Τα υποδείγματα αυτά δίνουν την δυνατότητα στις ε, χώρες ε, να τα μεταφράσουν αλλά και να τα τροποποιήσουν Ε, να βάλουν τα δικά του σήματα επάνω κτλ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προετοιμάζουμε μια έρευνα για την ετοιμότητα στις ε, χώρες, ε, συγκεκριμένα την ετοιμότητα των νοσοκομείων. Βεβαίω όλα αυτά δεν τα κάνουμε μόνοι μας. Είμαστε σε καθημερινή επαφή με την Γενική Διεύθυνση Υγείας, με το Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με τον αντίστοιχο φορέα στην ε, Κίνα και στη ΣΥΠΑ. Είμαστε σε επαφή και με τον αντίστοιχο φορέα στην Αφρική για να δούμε τις δυνατότητες και την ετοιμότητα που έχουν για να ανοιχνεύσουν περιπτώσεις ε, του κορονοϊού. Οπότε. Και τώρα τα χρειάζομαι την αξιολόγηση κινδύνου. Ε, ήθελα λίγο να συνοψίσω τις ε, δραστηριότητές μας με το πώς βλέπουμε τον κίνδυνο αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ο πιθανός αντίκτυπος ε, κρουσμάτων ε, του κορονοϊού είναι υψηλός. Η πιθανότητα μόλυνσης για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ ε, που κατοικούν ή επισκέπτονται την περιφέρεια αυτή Χουμπέη στην Κίνα είναι υψηλή. Η πιθανότητα μόλυνσης ε, σε άλλες κινέζικες περιφέρειες είναι μέτρια αυτή τη στιγμή, μπορεί να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες υπάρχει μια μέση ως υψηλή πιθανότητα να δούμε και άλλες, και άλλες αγόμενα κρούσματα και εάν τα κρούσματα ανοιχνευθούν νωρίς ε, και ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου της μόνσης, ε, ειδικά σε ε, κέντρα υγείας, η δυνατότητα περαιτέρω διάδοσης σε ανθρώπους εντός της Ένωσης θα είναι από χαμηλή ως πολύ χαμηλή. Εάν τα μέτρα αυτά δεν εφαρμοστούν και ανοιχτευτούν τα κρούσματα αργά, τότε βεβαίως ο κίνδυνος δευτερογενούς μετάδοσης ε, στην κοινότητα είναι υψηλός. Οπότε, ε, καταλήγω τώρα, ολοκληρώνω ε, για τον κορονοϊό. Θα μπορούσα βεβαίως να επεκταθώ και άλλο, αλλά φαντάζομαι θα μου κάνετε και ερωτήσεις. Θα ήθελα τώρα να φέρω κάποια παραδείγματα άλλων απειλών. Το ένα από αυτά είναι η, η Λάρα. Έχουμε 53.000 κρούσματα στην τελευταία, τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο είναι φτηνό και αποτελεσματικό. Αυτό οφείλεται εν μέρη στο ότι υπάρχει παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί Ε, και ανησυχεί ο κόσμος για το εμβόλιο. Γι' αυτό το 2018 έγιναν συστάσεις του Συμβουλίου ακριβώς για τις αρρώστιες οι οποίες προλαμβάνονται με εμβολιασμό και ως αποτέλεσμα αυτής της σύστασης το κέντρο μας αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται μια ευρωπαϊκή πύλη για τα εμβόλια, θα είναι πανευρωπαϊκή, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που θέλουμε να αποτελέσει την πηγή έγκυρων πληροφοριών για οποιονδήποτε θέλει να πληροφορηθεί σχετικά. Η πύλη αυτή θα ανέβει στα τέλη Απριλίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εμβολιασμού. Η άλλη απειλή ε, την ανέφερα ήδη είναι η αντίσταση των μικροβίων στα φάρμακα Μία από τις αξιολογήσεις κινδύνου που δημοσίευσαμε σήμερα αφορά ακριβώ κάποια κρούσματα στην ε, Λιθουανία και θα δημοσίευσουμε άλλη αυτή την εβδομάδα αφορά κρούσματα σε, πολλών, σε πολλές χώρες ε, του κολοβακτηριδίου το οποίο πλέον αντιστέκεται στα φάρμακα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι κάθε χρόνο γύρω στους 33.000 άνθρωποι πεθαίνουν ως αποτέλεσμα της αντίστασης ε, στα φάρμακα των ε, μικροβιών. Και αυτό συγκρίνεται με το βάρος ε, της γρήπης, της φυματίωσης και του HIV μαζί το βάρος στα συστήματα υγείας. Δηλαδή είναι μια αρκετά μεγάλη απειλή η οποία δεν απασχολεί τόσο πολύ τα ΜΜΕ όσο ο κορονοϊός. Ήθελα επίσης ε, να σας πω ότι κοιτάμε και εκτός της Ευρώπης για να προστατεύσουμε την Ευρώπη. Εδώ πέρα συνεργαζόμαστε είτε με τον ΠΟΕ είτε με τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και αυτή τη στιγμή ένας υπάλληλο μας βρίσκεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό όπου υπάρχει η επιθυμία της έμπολα η οποία δεν έχει ακόμα τελειώσει φαίνεται πως ε, πάει προς έλεγχο, αλλά ήδη έχει περάσει 1,5 χρόνος. Μετά θα ήθελα να τονίσω κάποια άλλα πράγματα που κάναμε το 2019, καθώς κάνουμε αυτή την ανασκόπηση. Συνολικά, πέρσι, βγάλαμε 23 ε, γρήγορες αξιολογήσεις κινδύνου, δεδομένου του ότι αυτή την εβδομάδα, αυτή, μέχρι τώρα έχουμε βγάλει ήδη 8, φαίνεται ότι το 2020 είναι κάπως πιο έντονο. Είχαμε 58 τεχνικές εκθέσεις για διάφορα θέματα, με διαβουλεύσεις, ε, γραπτά κοινοβουλευτικά ερωτήματα, όχι α, τόσα όσα συνήθως γιατί πέρσι είχαμε και τις εκλογές και δημοσιεύσαμε 86 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Ως προτεραιότητα φέτος, όπως είπα, έχουμε να δούμε το θέμα της αντίστασης ε, στα φάρμακα, το να δούμε την εφαρμογή των στάσεων του Συμβουλίου για την ενίσχυση της συνεργασίας για τις αρρώστιες που προλαμβάνονται με εμβόλια, να στηρίξουμε την Κομισιόν στο να επιτύχει τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικά όσον αφορά την ε, υπατήτηδα και τη φυματίωση και τον HIV. Ειδικά έχουμε τα θέματα της ηλεκτρονικής υγείας και εφαρμόζουμε και ένα πρόγραμμα πρόβλεψης όπου προσπαθούμε δηλαδή να προβλέψουμε κάποιες ε, μεταδοτικές ασθένειες που υπάρχουν ή θα έρθουν. Στηρίζουμε επίσης ε, τα κράτη-μέλη σε διασυνοριακές ε, περιπτώσεις ε, και εξετάζουμε και τους εσωτερικούς μας μηχανισμούς για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέτωπο της αποτελεσματικότητας. Τώρα, πέρα από δύο μήνες ενέκρινε το ΔΣ το πρόγραμμα μας για το 2020 γιατί βεβαίως οι περισσότεροι που μας εργαζόμαστε επί του κορονοϊού και θα παρουσιάσουμε κάποιες δραστηριότητες που θα κάνουμε. Τέλος, θα είχα να σας δείξω τις λέξεις κλειδιά για το έτος, δυστυχώς ούτε αυτό δεν μπορείτε να το δείτε. Ε, θα σας τη στείλουμε την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ, εν για την προσοχή σας. Now it's there. Πήρε μάλιστα. Start again. Άντε ξαναρχίστε τότε, αφού τις βρήκαμε τις διαφάνειες. Σας ευχαριστούμε κυρία μου. Ούτως ή άλλως θα σας στείλουμε την ε, παρουσίαση. Ως ονούπο, γιατί εγώ ως πρόεδρος έχω το προνόμιο και την έλαβα πρώτος και βλέπουμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, χάρτες και ούτω καθεξής, οπότε έχει νόημα να τη μοιράσουμε και όλα θα είναι πολύ ενδιαφέρον για του συναδέλφου. Και ίσω τι απαντήσεις μπορείτε να επανέλθετε σε κάποιε διαφάνειες και να τι ξανα... δείξετε. Ξεκινάμε με τους εκπροσώπους μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Όσων. Κυρία Κοπτσίνσκα πρώτη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Διευθύντρια, καλημέρα σας και πάλι. Έχουμε τακτικές επαφές και χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί για τον τακτικότατο διάλογο που έχουμε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Νόσων. Βέβαια, θα ήθελα αυτές οι συναντήσει να γίνονται σε διαφορετικέ περιστάσεις και για άλλους λόγους. Αυτή τη στιγμή δυστυχώ έχουμε επιδημιολογική απειλή, όπως έχει ανακηρύξει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ε, λόγω του κορονοϊού. Στις ε, συναντήσεις που είχαμε, η κυρία Διευθύντρια μας ενημέρωσε για το βαθμό ετοιμότητα των κρατών μελών στα πλαίσια τη ε, συνεργασία για την καταπολέμηση του ιού. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι κάποιε χώρε μέλη ε, πρόσφεραν βοήθεια για την ε, επεξεργασία διαγνωστικών και εργαστηριακών τεστ σε περίπτωση που κάποιες χώρες ε, ζητήσουν διάγνωση για ανθρώπους που είναι ύποπτοι να φέρουν τον ιό. Επίσης, μα μας θύμισε την επιδημία του ΣΑΡΣ του 2003 και του ΜΕΡΣ του 2012 η κυρία Διευθυντρία και τις και την αντιμετώπιση που είχαμε τώρα. Ελπίζω να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και τον νέο κορονοϊό και να κρατήσουμε την επαγρύπνησή μας. Τώρα, το ECDC, που είναι εκτελεστικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να προσφέρει βοήθεια προκειμένου να έχουμε συντονισμένες ενέργειες και ενιαία ε, προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ε, διάγνωση του κορονοϊού στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε. Ε, Στου υπηκόου ή στους διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και μη Ευρωπαίου υπηκόους. Σε περίπτωση που αρχίσει να μεταδίδεται ο ιός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα συστήσει το ECDC στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ανοιχνευθούν οι φορείς και το, το στενό του περιβάλλον και πώ ε, θα έχουμε το συντομότερο δυνατό ε, διαγνωστικά τεστ και με ποιο τρόπο. Επίσης, σε σχέση με τη συνεργασία με το κέντρο λιμωδών. Έχετε άμεσες επαφές με το κέντρο αυτό ή ε, μέσω μόνο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ή κάποιους διεθνείς φορείς. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε θερμότατα για τις ασθενές ε, και πολύ τακτικές επαφές που έχετε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Ε, μέσα σε μία ομιλία διατυπώσατε 4-5 ερωτήσεις. Οπότε ας ξεκινήσουμε με τις απαντήσεις. Κυρία Διευθύντρια, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Η ερώτηση για, τους, ε, για την εργαστηριακή υποστήριξη και τα διαγνωστικά τεστ. Όντως, κάποιες χώρες πρόσφεραν ε, να ελέγξουν ε, δείγματα από άλλες χώρες. Σε περίπτωση όμως που δεν έχουμε τόσο μεμονωμένα κρούσματα όπως τώρα, αλλά μια μεγαλύτερη εξάπλωση ε, της νόσου ή του ιού, σε τέτοια περίπτωση δεν χρειάζεται να γίνεται διάγνωση κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. Γιατί κάτι τέτοιο θα κατακλείσει ε, τα εργαστήρια με τεράστιο αριθμό ε, αιτήσεων. Θα πρέπει όμως να βρούμε έναν αλγόριθμο για να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της έξαρσης και της εξάπλωσης του ιού στα κρατημέλη χωρίς να χρειάζεται να ελέγχουμε κάθε φορέα ή κάθε ύποπτο ε, για το κρούσμα. Πάντως, αν έχουμε συγκεκριμένες αιστείες, δεν μπορούμε να ελέγχουμε τους πάντες. Όταν έχουμε πανδημία δεν κάνουμε μεμονωμένες ανιχνεύσεις, γιατί σε ομάδες με παρόμοια συμπτώματα, αρκεί να γίνεται διάγνωση σε έναν. Υποθέτουμε ότι οι υπόλοιποι που φέρουν τα ίδια συμπτώματα πάσχουν από την ίδια νόσο. Δεν χρειάζεται να ελέγχουμε τον καθένα ξεχωριστά. Θα δούμε όμως πώς θα ενεργοποιήσουμε αυτούς τους πόρους, ώστε να κάνουμε σωστή αξιολόγηση των πόρων. Σε ό,τι αφορά το Κινέζικο Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, έχουμε συνεργασία με το Κινέζικο Κέντρο πρόληψης και ελέγχου νόσων. Έχουμε τακτικές επαφές. Έχουμε λάβει και τη μεταφρασμένη ε, έκθεσή τους ε, για την κατάσταση του ιού. Και σίγουρα οι συνάδελφοι εκεί υφίστανται τεράστιες πιέσεις. Έχουμε την αίσθηση πάντως ότι πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν για να μας κοινοποιήσουν τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. Μάλιστα, περνάμε στο Catch the Eye τώρα. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο των ομιλητών. Mr. Sadas, Véronique Rielenoir, Azekamp, Mr. Wallace, Srivasi, TMS, one more, two more, three more, over. The next one will cost a lot of points. Έχουμε το κατάλογο τον κλείσαμε. 1,5 λεπτό καθένας παρακαλώ με ερωτήσεις μόνο για να προλάβει η διευθύντρια να απαντήσει διεξοδικά. Ξεκινάμε τον Πέτερ Λίζε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε και να μιλήσω. Πράγματι το θέμα είναι ενισχυτικό, πολλοί άνθρωποι ανησυχούν και βεβαίω εντάξει γεγονό είναι πως υπάρχουν πολύ περισσότεροι θάνατοι από άλλες ασθένειες. Ε, αναφέρατε την αντοχή στα αντιβιωτικά, τη μικροβιακή αντοχή και ε, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε ενήμεροι και σας ευχαριστώ για τις ε, πληροφορίες. Θεωρώ ότι τώρα η δικιά μας η δουλειά είναι να μην δημιουργήσουμε πανικό, να καθισχάσουμε τον κόσμο. Βεβαίως ε, υπάρχουν, όπως είπατε, και επαφέ με τη Γουχάν. Ε, δύο ερωτήματα έχω. Θα μπορούμε να περιμένουμε μετάλλαξη του ιού ή θεωρείτε πως είναι απίθανο. Δεύτερον, υπάρχουν σοβαροί επιστήμονες που λένε πως οι κινέζικες αρχές ε, δεν μας λένε τους πραγματικούς αριθμούς και έχουν διάφορες ενδείξεις ε, με βάση τα όσα διαπιστώνουν στην Ευρώπη και σε άλλα σημεία του πλανήτη ή θεωρείτε ότι ε, είμαστε ενημερωμένοι σωστά. Κυρία Γιώτελαντ, για το S&D. Ευχαριστούμε την κυρία Άμον, ευχαριστώ πρόεδρε, που βρίσκεται εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε αυτά τα πολύ χρήσιμα στοιχεία όχι μόνο τις ε, οξύες κρίσεις δηλαδή που αντιμετωπίζουμε αλλά και τα πιο μακροπρόθεσμα προβλήματα. Είναι πολύτιμη η εμπειρία που έχετε συλλέξει, που έχουμε συλλέξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που μας κάνει πλέον ασφαλέστερους. Και μιλώ για το SARS, μιλώ για τις εμπειρίες που έχουμε αφήσει πλέον πίσω μας αισθανόμαστε ασφαλέστεροι που αυτά, αυτό το πεδίο καλύπτεται πλέον από το κέντρο σας. Συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή ότι δεν πρέπει να σπείρουμε τον πανικό, πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί, να παρακολουθούμε την κατάσταση, να ανταλλάζουμε βέλτιστες πρακτικές με τα κράτη-μέλη, να προστατεύουμε τους πολίτε μα από τη μετάδοση οποιοδήποτε ιού ή νοσήματος. Και γι' αυτό πολύ χαίρομαι που συνεργάζεστε με τον ΠΟΗ όπως μας είπατε. Εγώ έχω μια ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, όταν έρχονται άνθρωποι από την Κίνα, ε, αναρωτιέται πολλοί κόσμος κατά πόσον μπορούν να μεταδίδουν, να μεταδώσουν την όσο. Πώς μπορεί να προστατευθεί κανείς από τη μετάδοση, από τα συμπτώματα. Αλλά δεύτερη ερώτηση, ακριβώς αν έχει κανείς προσληφθεί από τον ιό. αν κάποιος έχει συναντήσει κάποιον άλλο άνθρωπο που ίσως να μην πρόσεχε τόσο πολύ, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η δεύτερη γενιά μετάδοσης, για να το πω έτσι, οι άνθρωποι που ήδη βρίσκονται στις χώρες μας, θα γνωρίσουν καλύτερα τα συμπτώματα ώστε να αντιληφθούν ότι έχουν προσληφθεί. Και πολύ χαίρομαι που αναφερθήκατε και στην Ιλαρά και στα θέμα της μικροβιακής αντοχής που ανέφεραν και άλλοι ομιλητές. Πιστεύω ότι πρέπει να εστιαστούμε ιδιαίτερα σε αυτό και θα ήθελα να ξέρω από εσά τι επιθυμείτε, τι χρειάζεστε εσύ από εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Νουάχ από το Ρινιού, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ την Διευθύντρια. Η επιδημία αυτή μας δείχνει πόσο διεθνής είναι η κίνδυνη για την υγεία, πόσο χρειάζεται συλλογική αντιμετώπιση, δεν γνωρίζουν σύνορα οι ΙΕΙΣ οι λύσει μόνο παγκόσμιες, διεθνεί ή εν πάση μπορεί να είναι. Εγώ χαιρετίζω τις δράσεις σα ε, και τον συντονισμό και την παρακολούθηση. Ως ιατρός εγώ παρακολουθώ καθημερινά τις ε, αρχές ε, της δημόσιας υγείας στη χώρα μου, τις συστάσεις του ΠΟΗ που απευθύνονται στους επαγγελματίες της υγείας ώστε να εντοπίσουμε και να ε, φροντίσουμε τους ανθρώπους που έχουν προσληφθεί. Διερωτώμε όμως για την υλοποίηση των συστάσεων αυτών στις διάφορες χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα στις χώρες που κυρίως ενέχονται. Γιατί ως προς τις μεταδοτικές νόσους ε, δεν έχει νόημα να λαμβάνουμε οποιοδήποτε μέτρο αν δεν είναι να το λαμβάνουμε όλοι παντού στον κόσμο. Επομένως ως προς την υλοποίηση των συστάσεων του ΠΟΗ τι θα είχατε να μας πείτε κυρία Διευθύντρια, ιδιαίτερα στο κινέζικο έδαφος, στην κινέζικη επικράτεια. Πρόεδρος, να ακούσουμε άλλες τρεις ερωτήσεις αν συμφωνείτε, κυρία Διευθύντρια, και θα σας δώσω το λόγο. ID, παρακαλώ. Ε, κυρία Διευθύντρια, αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια απειλή για την ε, δημόσια υγεία με την εξάπλωση του κορονοϊού. Η εξέλιξη είναι ταχύτατη και ίσως μπορεί να εξελιχθεί αυτή η επιδημία σε πανδημία. Σε αυτό το πλαίσιο οι πολιτικές μετανάστευσης και ε, ελέγχων στα σύνορα διευκολύνουν φοβούμε, λυπούμε που το λέω, την εξάπλωση του ιού αυτού και της νόσου αυτής. Ιδιαίτερα μιλώ για τους αερολιμένες, αλλά και τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα, που μπορεί να τα περάσει κανείς με μεγάλη ευκολία. Είχαμε συζητήσει και πρόσφατα το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων για Κινέζους πολίτες. Ε, στο πλαίσιο αυτό η μετάδοση των ιών δεν θα πρέπει να εξωθήσει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ξαναδούν, να επαναξετάσουν τις πολιτικές ε, ε, μετανάστευσης που εφαρμόζουν και το πλαίσιο του Σέγγεν και τα, τους έλεγχους στα σύνορα. Η πράσινη παρακαλώ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Δευθύντρια. Κοιτάξτε, εγώ Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά για τον κορονοϊό. Δεν ξέρω αν έχετε ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη στη διάθεσή σα. Δηλαδή, γνωρίζουμε από πού έρχεται. Αρχικά είχαν πει για τις νυχτερίδες, μετά είχαν πει για άλλα πράγματα. Τι γνωρίζετε για, το, για την προέλευσή του. Επίσης για τις δυνατότητε μετάλλαξης αυτού του ιού. Έχετε κάνει γενετική ανάλυση, γενετικές δοκιμές από τα δείγματα από την Κίνα, είχαμε και στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν έχει ήδη γίνει η μετάλλαξη του ιού. Επίσης για την μεταδοτικότητά του έχουμε ανθρώπους που ήρθαν στη Γαλλία, βρίσκονται δύο εβδομάδες τώρα σε καραντίνα. Ε, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσος χρόνος χρειάζεται. Επίσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ στην Ευρώπη έχουμε τις δομές της δημόσιας υγείας για να φροντίσουμε τους ασθενείς. Αλλά στην Αφρική, στην Καραϊβική, αν εκεί έχουμε κρούσματα μετάδοσης, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχετε μήπως συγκεκριμένες πληροφορίες και για τη διάγνωση. Γιατί μας λέτε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πλήρη διάγνωση για να γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια απλή γρήπη ή για συμπτώματα του ιού. Και επ' αυτού θα ήθελα να ακούσουμε τις συστάσεις σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ για τον πρώτο γύρο η κυρία Αζεκό. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις για τη χρήση των αντιβιωτικών στην ε, κτηνιατρική και στην κτηνοτροφία, αλλά θα περιοριστώ στον κορονοϊό. Σύμφωνα με το Reuters φαίνεται ότι τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν στο Γουχάν μέσω ζώων μεταξύ των οποίων λύκη φίδια, νυχτερίδες και τα λοιπά. Οπότε το ίδιο φαίνεται ότι συνέβη και με το SARS το οποίο μεταδόθηκε από τα άγρια ζώα στον άνθρωπο και αυτός ο ιός ξεκίνησε από την Κίνα και ο ιός Μέρς επίσης μεταδόθηκε από τα ζώα στον ε, άνθρωπο. Μήπως το να σταματήσουμε να εμπορευόμαστε και να τρώμε ε, άγρια ζώα θα βοηθούσε την... το να μην μεταδοθεί ξανά ένας τέτοιος ε, ιός τουλάχιστον να σταματήσουμε να τα εισάγουμε από την Κίνα. Νομίζω θα είναι καλό για τους ανθρώπους και οπωσδήποτε για τα ζώα. Thank you. <laughs> Easy ones. Yeah, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πολύ άριθμες ερωτήσεις σας. Καλύψετε ένα ευρύτατο φάσμα. για να δούμε για, το δυναμικό μετάλλαξης του νέου κορονοϊού. Δύο ευρωβουλευτές έθεσαν την ίδια ερώτηση. Όντως, οι «ή» μεταλλάσσονται. Μεταλλάσσονται με διαφορετική συχνότητα βέβαια. Σε ό,τι αφορά αυτό το νέο κορονοϊό, δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες για τη δυνατότητα μετάλλαξης ή την ταχύτητα ή συχνότητα μετάλλαξης. Φαίνεται σαν να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό εδώ και πολύ καιρό, αλλά σκεφτείτε ότι μόλις πριν τρεις εβδομάδες ε, ουσιαστικά εντοπίστηκε αυτός ο νέος κορονοϊός. Οπότε είναι λογικό να έχουν μείνει ακόμη αναπάντητα πολλά ερωτήματα. Ίσως σε λίγες εβδομάδες από τώρα θα έχουμε και άλλες απαντήσεις, αλλά ακόμη δεν τις έχουμε όλες. Και σίγουρα δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα για την δυνατότητα μετάλλαξης του ιού. Σίγουρα όμως ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα κάποια στιγμή. Γιατί η μετάλλαξη του ιού θα επηρε... επηρεάσει και τη διάγνωση στο εργαστήριο και τη θεραπεία μεταγενέστερα του ιού. Πολύ σημαντική ερώτηση, αλλά δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε απάντηση. Επίσης, αν είναι σωστά τα στοιχεία που μας δίνει η Κίνα για τα κρούσματα και τους νεκρούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε υποψίες για το ότι μας δίνει ανακριβή στοιχεία. Και μάλιστα είδαμε ότι τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες 7 με 10 μέρες, περάσαμε από 1.200 νέα κρούσματα τη μέρα σε 2.800 κρούσματα τη μέρα, όπως μάθαμε χθες και σήμερα. Αυτή η μεγάλη αύξηση δείχνει κατά τη γνώμη μου ότι υπάρχει καλύτερη διάγνωση, όχι κατά ανάγκη ότι πριν μας απέκριμα στοιχεία, για να απαντήσω την ερώτηση, στην ερώτησή σας λοιπόν ξεκάθαρα, μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξει ότι η Κίνα αποκρύπτει κάποια στοιχεία. Αλλά ακόμη και το έκανε δεν θα το μαθαίναμε. Ε, σαφέστατο. Δεν βοηθάει, το ξέρω. Αλλά μόνο πληροφορίες που έχουμε μπορούμε να εξετάσουμε και να σχολιάσουμε. Και η οικοτολογία αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει. Εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση και αν διαπιστώσουμε διαφορές μεταξύ των στοιχείων που μας δίνει η Κίνα και άλλων που συγκεντρώνουμε, θα το θέσουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα ύποπτο πάντως, ή αμφισβητήσιμο. Ρωτήσατε τι θα κάνουμε με τον κόσμο που έρχεται σε ευρωπαϊκές χώρες ε, από την Κίνα. Σε τελική ανάλυση αυτό αποτελεί ευθύνη των εθνικών αρχών υγείας, των εθνικών υγειονομικών υπηρεσιών. Αυτό που κάναμε, δεν μπορώ να σας το δείξω δυστυχώς, είναι ότι συντάξαμε ένα έντυπο ενημερωτικό στο οποίο αναφέρουμε τι θα πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες που έρχονται από την Κίνα. Για παράδειγμα, αν έχουν σύμπτωμα λίμωξης του αναπνευστικού συστήματος, θα πρέπει να αποτανθούν σε ένα γενικό παθολόγο ή να πάνε σε ένα νοσοκομείο ή στον αρμόδιο φορέα και να παρουσιάσουν, όχι μόνο, να περιγράψουν όχι μόνο τα συμπτώματά τους, αλλά να πούν και το ιστορικό το, του ταξιδιού τους. Γιατί αυτή την εποχή του χρόνου τέτοια συμπτώματα του αναπνευστικού είναι συχνότατα. Οποιοςδήποτε έχει κρύωμα δεν μπορεί να ελέγχεται για τον κορονοϊό. Αν έπρεπε να ελέγξουμε το κάθε κρύο με την κάθε γρήπη, θα κατακλείζονταν τα εργαστήρια και δεν θα οδηγούμασταν πουθενά. Οπότε θα πρέπει να αναφέρεται πότε έγινε το ταξίδι και σε ποια περιοχή της Κίνας. Αυτή είναι η σύσταση που αναφέρουμε στο ενημερωτικό φυλάδιο που συντάξαμε. Τώρα, αν θα λάβουν τις δικές μας συστάσεις οι χώρες ή θα συντάξουν δικά τους ενημερωτικά φυλάδια, αυτό είναι δική τους ε, δουλειά. Πάντως εμείς έχουμε ήδη δημοσιεύσει συστάσεις. Ρωτήσατε επίσης ε, αν ε, μπορούμε να υπολογίσουμε κατά πόσο εκείνη εφαρμόζει τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όχι, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Είναι κάτι που μπορούμε να ρωτήσουμε βέβαια. Και θα το φροντίσω, θα δω τι ενημέρωση υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΠΟΗ για το κατά πόσο εκείνη εφαρμόζει τις συστάσεις του. Δεν ε, είμαστε εμείς αρμόδιοι να το ελέγξουμε, μπορούμε όμως να το ρωτήσουμε στους συναδέλφους ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επίσης, ε, μια έκκληση προς σε εμάς και τις, να συστήσουμε στις χώρες να διακόψουν το χώρο Σέγγεν. Εμείς είμαστε επιστημονικός φορέας, επιστημονικό κέντρο. Δεν είμαστε πολιτικό όργανο, ούτε μπορούμε να λάβουμε τέτοιες αποφάσεις αναστολής του Σέγγεν. Από επιστημονική άποψη πάντως στην Ευρώπη δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αναστολή του χώρου Σέγγεν. Από πού προήλθε ο ιός. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και όλοι θυμούνται ότι στην αρχή είχαμε πει ότι όλα τα κρούσματα έχουν σχέση με αυτή την αγορά ζώων του Βουχάν. Όπως είπατε και οι προηγούμενοι κορονοϊού είχαν κάποια σχέση, μερικοί έστω, ε, ή κάποιο δεσμό με ζώα, μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο. Και ήταν αρκετά αληθοφανής ε, αυτή η προέλευση. Μετά όμω ε, προέκυψε μετα ομως προεκυψε οτι δεν ήταν αδύνατο να είναι μόνος, ο μόνος τρόπος μετάδοσης. Γιατί μόνο από, τις από τα πολλά αρχικά κρούσματα μόνο 100 είχαν άμεση επαφή με ζώο. Οπότε στην αρχή μπορεί να ήταν δυνατή μετάδοση από ζώο, αλλά στη συνέχεια ο ιός μεταδόταν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και αυτό φάνηκε πολύ γρήγορα. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Κίνα είναι εμφανώς μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν χρειάζεται πια να μεσολαβούν ζώα. Τώρα, περίοδος επόασης του ιού. Και αυτό το μαθαίνουμε εν το γίγνεσθε στην πορεία όσο περνάει η ώρα. Ο χρόνος επόασης αυτή τη στιγμή υπολογίζεται σε 3 με 12,5 μέρες. Οπότε σε αυτήν την απομόνωση στην καραντίνα έχουμε προβλέψει 14 ημέρες σε περίπτωση που είναι κάπως μεγαλύτερος ο χρόνος επόασης θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος. Αν το διαπιστώσουμε θα προσαρμόσουμε την καραντίνα, γιατί κάποιοι έχουν χρόνο επόεσης τρεις εβδομάδες. Πάντως θα δούμε ανάλογα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε πώς θα προσαρμόσουμε τις συστάσεις μας. Τώρα για τις χώρες ΑΚΕ. Όντως έχετε δίκιο και γι' αυτό έχουμε επαφές με το Αφρικανικό Κέντρο Λιμωδών Νόσων Δυστυχώ δεν μπορούσα να σας δείξω το χάρτη, αλλά μέχρι στιγμής στην Αφρική δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα. Πάντως έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με το Αφρικανικό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αν χρειαστεί και αν μπορούμε. Κυρία Χάζεκαμπ, ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση σας για το εμπόριο με τα άγρια ζώα ή την απαγόρευση. Δεν νομίζω ότι θα βοηθούσε κάτι τέτοιο τώρα. Δεν λέω ότι δεν είναι λόγος ε, κάποια στιγμή να σταματήσει, αλλά όχι, δεν θα, η απαγόρευση του εμπορίου αγρίων ζώων αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επηρεάσει την περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού. Τώρα, για τις ερωτήσεις που δεν αφορούν τον κορονοϊό, ας τις αφήσουμε για τον τελευταίο γύρο. Κυρία Ευχαριστώ τη Διευθύντρια που ήρθε εδώ και μας εξήγησε πώς έχει εικόνα σχετικά με τον ιό αυτό. Ε, με ενδιαφέρει και το τελευταίο τμήμα της τοποθέτησής σας για άλλες περιπτώσεις ε, νόσων και την ικανότητα του κέντρου και των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν τις νόσεις αυτούς, γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο ε, γρήπης ε, και της Ιλαράς πώς έχουν εδώ οι δυνατότητες μας, πώς θα πάμε. Επίσης, ποια είναι η σχέση μεταξύ της Κίνας και ε, του ECDC και του ΠΟΗ και δεν ξέρω αν εμπίπτει αυτό στο πεδίο σας, αλλά γνωρίζετε κατά πόσον ο ΠΟΗ έχει κάποιον επιτόπου στην Κίνα, έχει κάποιον σύνδεσμο για να επιβεβαιώσουμε ενδεχομένως τους, ε, τον βαθμό θνησιμότητας που μας έχει διαβιβαστεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Πόλτσα και το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για την μικροβιακή αντοχή. Διότι Πρόκειται για μια συζήτηση, ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον και αφορά και άμεσα και την ε, κοινή γνώμη. Διότι εγώ εξεπλάγινα από τις ε, χιλιάδες θυμάτων που ακούσαμε ότι υπάρχουν. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να διαβιβάσουμε καλύτερη ενημέρωση, καλύτερες πληροφορίες στους πολίτες μας, να εξηγήσει η Επιτροπή στους πολίτες τι σημαίνει μικροβιακή αντοχή και τι στάση πρέπει να τηρούν οι πολίτες ώστε να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόρβαλς για το Ρινιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Άμον που είναι εδώ μαζί μας. Ίσως έπρεπε να έχουμε την Μαρλέν Ντίτριχ ε, στο... από πίσω να μας τραγουδάει ε, πότε θα καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι. Ε, γιατί είχαμε και ένα άρθρο στο New York Times για έναν οφθαλμολόγο που είχε προσπαθήσει να προειδοποιήσει αλλά του έκαναν παρατήρηση. Δηλαδή Ίσως εδώ να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το απολυταρχικό κινέζικο κράτος προσπαθεί να περιορίσει την ενημέρωση και την πληροφορία και ίσως και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διαβάσουμε στον ΠΟΗ. Γιατί πρόκειται για θανάσιμη παγίδα. Αυτό το απολυταρχικό καθιστός δηλαδή είναι η θανάσιμη παγίδα. Μάλιστα. Ε, S&D παρακαλώ. Ο κύριος ε, Κασάρες, ευχαριστώ, πρόεδρε, ευχαριστώ την ε, διευθύντρια που είναι εδώ σήμερα και μας μιλάει για το πολύ σημαντικό θέμα του κορονοϊού, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πανικό που επικρατεί. Ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας, την ευφυΐα μας, τα μέσα που διαθέτουμε σε πλαίσια δημόσιας υγείας, ώστε να αντιμετωπίσουμε το SARS, την γρήπη Α, τον έμπολα, οποιαδήποτε άλλη απειλή, οποιοδήποτε άλλον κίνδυνο. Το να κυκλοφορούν φήμες ότι πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα, ότι πρέπει να αναστείλουμε το Σέγγεν και όλα αυτά, μου φαίνονται ανεύθυνα ε, χωρίς να έχουμε και πολύ συγκεκριμένες και αξιόπιστες πληροφορίες. Όλα αυτά δεν θα συνεισέφεραν μάλιστα και σε τίποτα. Απλώς ε, τρέφουν λαϊκισμούς ε, και κινδυνολογίες για καταστροφικές συνέπειες οι οποίες στην ουσία δεν επιβεβαιώνονται. Από τα όσα γνωρίζουμε για τα εργαστηριακά μέσα, πότε, πότε νομίζετε, πότε θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε έναν αλγόριθμο που θα μπορούσε ίσως να μας βοηθήσει στην ε, διάγνωση. Και από ό,τι φαίνεται η μετάδοση του ιού γίνεται μέσω του αναπνευστικού και οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, τα πιο ε, σοβαρά κρούσματα ε, διαγιγνώσκονται μέσω του πρωτοκόλλου Μούρστα, αν ακούσαμε καλά την ομιλητή. Αυτό δεν θα μπορούσε να μας βοηθήσει στις πιο σοβαρές αυτές περιπτώσεις. Επίσης, ε, οι ασθενείς, τα θύματα αυτά ή οι πιο σοβαρές περιπτώσεις ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές αγωγές αντιστοίχων νόσων. Και επίσης, μιλούμε για τον νόσο αυτή, μιλούμε για τον ιό, αλλά στην Αφρική, στο Κονγκό, έχουμε άνω των 3.000 ασθενών και άνω των 2.000 νεκρών από τον έμπολα. Επομένως, ποιες είναι οι προγνώσεις ή οι προβολές σχετικά με τον έλεγχο, τον περιορισμό του έμπολα στην Αφρική. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Μόνο για την εξήγηση που μας έδωσε. Εγώ ήθελα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι φαντάζομαι, να καταλάβω τι κάνει το ECDC για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Μας δώσατε εξηγήσει. Εγώ εξ όσων γνωρίζω ε, προήλθε από παράνομη αγορά κρέατος, ο ιός αυτός λέει ο Οπότε ήθελα να σας ρωτήσω για την ε, ρύθμιση της αργοράς αγρίων ζώων στην Ευρώπη, διότι έχουμε περιπτώσεις που μας δείχνουν ότι οι εισαγωγές κρέατος στην Ευρώπη, που είναι 270, 270 τόνοι το χρόνο, εκτός από το, το πλήγμα στην βιοπικιλότητα, με συγχωρείτε, μπορεί να είναι και πηγή διαφόρων νόσων που επεκτείνονται παντού στον κόσμο. Μετά την κρίση έμπολα και την ε, μετάδοση ε, η ΕΦΣΑ αναγνώρισε σχετικά με τις ε, παράνομες αυτές τις αγωγές ότι υπήρχε πραγματική απειλή για την δημόσια υγεία από τις αγωγές αυτές. Επομένως, η διεθνής λαθρεμπορία είναι μια υπαρκτή πηγή προέλευση ε, απειλών και κινδύνου. Ποιες δράσεις έχουν αναλυφθεί για να βελτιωθούν οι έλεγχοι και να σταματήσουν αυτές οι παράνομες εισαγωγές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γουάλλας για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για τον ε, κορονοϊό. Ε, ως προς την διαφάνεια της έκρηξης και των στοιχείων των δεδομένων που έχουμε στην ε, διάθεσή μας, την έγκαιρη διάγνωση, την απομόνωση, την καρατίντα και την οικοδόμηση των δύο νοσηλευτικών κέντρων, εσείς θεωρείτε ότι η κινέζικη κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί, έχει, λαμβάνει επαρκή μέτρα. Δεύτερον, εξεφράστη μια ανησυχία στην Ιρλανδία για μια πτήση από την Μόσχα, όπου υπήρχε ένας Κινέζος υπήκος που ασθενούσε στο αεροσκάφος. Μετά την προσγείωση κράτησαν το αεροσκάφος για δύο, χρόνιες, ε, για δύο ώρες, με συγχωρείτε, απομακρύνθηκε ο άνθρωπος αυτός και μετά ανακάλυψαν οι ιατροί ότι δεν είχε, δεν ασθενούσε από τον ιό. Όμως οι υπόλοιποι επιβάτες τους επιτράπει να αποχωρήσουν κανονικά. Αυτό είναι κανονικό είναι σωστή η εφαρμογή δηλαδή κάποιου μέτρου. Δεν έχουμε επικαιροποίηση και των ιστοσελίδων των ε, δημοσίων αρχών στην Ιρλανδία. Δεν έχουμε κατάλογο ε, κρουσμάτων ή περιπτώσεων. Δεν έχουμε τοποθεσίες. Εσείς συνεργάζεστε λοιπόν με τα κράτη-μέλη γιατί μιλάτε για ενημερωτικά φυλάδιο. Ε, εγώ αναρωτιέμαι τι οδηγίες, συστάσεις, συμβουλές έχετε δώσει στις αρμόδιες αρχές τα κράτη-μέλη όπως στη χώρα μου, στην Ιρλανδία. Σε τέτοιες αυτές συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως σας ανέφερα για την πτήση και δεν κινδυνολογώ, ε, ε, τι, πρέπει, τι μέτρα πρέπει να αναλαμβάνουν οι αρχές και είναι σωστά αυτά που έχουν κάνει μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ λέει Άρα, η κυρία Άμον έχει 10 λεπτά στη διάθεσή της για να απαντήσει σχετικά με τον ε, κορονοϊό και τις υπόλοιπες ερωτήσεις που έγιναν. Ωραία. Το ερώτημα ήταν ε, πώς επηρεάζει ο κορονοϊός τις δυνατότητές μας ε, για τα υπόλοιπα. Αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα αυτή τη στιγμή πέντε χώρες ε, επηρεάζονται και βεβαίως αφιερώνουν πολλούς ε, πόρους ε, σε αυτό. Υποθέτω ότι συνεχίζεται η παρακολούθηση και των άλλων ασθενειών, αλλά υπάρξει επιδημία, ίσως φτάσουν στα όρια τους. Αν μας ζητηθεί βεβαίως μπορούμε να στηρίξουμε, αλλά ε, η δική μας η δυνατότητα είναι και αυτή περιορισμένη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ε, δώσουμε κι εμείς κάποιες προτεραιότητες και στις ε, χώρες ε, στο τι κάνουμε. Ε, να επιβεβαιώσω επίσης ότι επικοινωνούμε απευθείας με τους ομολόγους μας στην Κίνα, όχι μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και έχουμε προβλέψει ακριβώς να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και είχε γίνει αυτό, παραδείγματο χάρη, στην περίπτωση της γρήπης των πτηνών που είχαμε εκεί και υποθέτω ότι ο έχει προσωπικό εκεί. Υπάρχει ένα περιφερειακό γραφείο νομίζω στη Μανίλα και αρκετοί από τους επιδημιολόγους που εκπαιδεύονται είναι έτοιμοι να μεταβούν εκεί. Για την ε, μικροβιακή αντοχή. Ναι, πράγματι, ο κόσμος πρέπει να ξέρει και κάθε χρόνο από το 2008 έχουμε μία μέρα και μία εβδομάδα ολόκληρη όπου αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα και προς ε, το ευρύ κοινό αλλά και για τους επαγγελματίες της υγείας γιατί ε, για να περιοριστεί ακριβώς η μικροβιακή αντοχή. Όλοι έχουν ένα ρόλο να παίξουν. Οι ασθενείς, οι γιατροί, οι αρχές, οι υγειονομικές, οι πολιτικοί, οι κτηνίατροι, οι οδοντίατροι, όλοι. Λοιπόν, ε, οι εξαιρετίες αυτές κάθε χρόνο απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο φάσμα όπου λέμε ε, τώρα είναι ευθύνη σας το θέμα αυτό. Γίνεται λοιπόν, βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες για κάποιους από τους παθογόνους παράγοντες υπάρχει μια σταθεροποίηση, για άλλους ακόμα και μείωση, οπότε υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει η κατάσταση και ε, βέβαια συμβαίνει αυτό. Μετά. Το γεγονός ότι οι Κινέζοι λαμβάνουν ε, αυστηρά μέτρα. Ε, είναι κάτι το οποίο δεν ε, λειτουργεί παντού. Αμφιβάλλω ας πούμε ότι ε, κάτι σαν αυτό το οποίο συνέβη στο Ουχάν μπορεί να γίνει στην Ευρώπη να λειτουργήσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως αυτομάτως ότι σημαίνει αυτό ότι κρύβουν πληροφορίες. Κοιτάξτε, έχει ασκηθεί δρυμία κριτική στην Κίνα μετά το SARS και νομίζω ότι έχουν διδαχτεί πλέον όσον αφορά ακριβώς ε, τις πληροφορίες ε, και ε, νομίζω έδωσαν τις πληροφορίες πάρα πολύ γρήγορα και για το στέλεχος. Είναι διαφορετική η κατάσταση από ό,τι πριν από 15 χρόνια. Μετά. Ένας αλγόριθμος Αν κατάλαβα καλά, ρωτήσατε και για το πόσοι ακριβώς ασθενούν από σοβαρές ε, αρρώστιες. Ε, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές ε, βεβαίως η μόνηση είναι ήπια. υπάρχουν και σοβαρές περιπτώσεις και θάνατοι και η θνησιμότητα θα έλεγα είναι ακόμα χαμηλότερη από ό,τι για τον SARS, αν και πρέπει να είμαστε ε, προσεκτικοί, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τη θεραπεία, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, κάποια συγκεκριμένη θεραπεία. Συμπτωματική είναι τα συμπτώματα, δηλαδή και όταν είναι πιο βαριά αυτά, αλλά Υπάρχουν βεβαίως ε, κάποια πειράματα που γίνονται για να δούμε αν κάποια αντιγυγικά θα μπορούσαν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα και όσον αφορά το Κόγκο. αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται κάθε εβδομάδα μειώνονται σταδιακά και όπως γνωρίζετε ε, υπάρχει εκεί πέρα και εμφύλιος πόλεμος οπότε οποιαδήποτε δυσκολία στον ε, τομέα της ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση της επιδημίας. Οπότε ε, φαίνεται τέλος πάντων ότι σταδιακά μειώνεται. Τώρα, όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει η παράνομη εισαγωγή κρέατος ε, ε, σφαγμένου στη ζούγκλα κτλ. Εκεί πέρα δεν μπορώ να σας δώσω κάποια απάντηση. Όπως λέτε αυτό περισσότερο αφορά την ΕΦΣΑ και την Κομισιόν. Ναι, για την Ιρλανδία. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη με αυτό το αεροπλάνο αλλά το γεγονός ότι οι άλλοι επιβάτες έφυγαν, δεν ξέρω αν τους άφησαν απλά να φύγουν, ε, σίγουρα θα έδωσαν τα στοιχεία τους για να μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους οι υγειονομικές αρχές. Όσον αφορά το πώς ε, χειρίστηκαν τις ε, πληροφορίες. Αυτό είναι κάτι που αποφασίζουν οι εθνικές αρχές. Εμείς μπορούμε απλά να διαθέσουμε τις δικές μας πληροφορίες ε, και έχουμε έναν μηχανισμό από το 2013 όπου οι χώρες ανταλλάσσουν πληροφορίες για το τι κάνουν τι μέτρα εφαρμόζουν και εκεί έχουμε λάβει διάφορες πληροφορίες. Τώρα δεν μπορώ, δεν θυμάμαι για την Ιρλανδία. Αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν κάποια μέτρα για να ενημερώσουν τον κόσμο. Αυτά νομίζω. Νομίζω απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σα ευχαριστώ σε 8 λεπτά. Να συνεχίσω. Μάλιστα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, θα δώσω το λόγο και στους δύο εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου, Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Όσων, στην κυρία Κούιοβιτς και στην κυρία Κοπάπο, δύο λεπτά η καθεμία. Ευχαριστώ κύριε Καμφά, κύριε Πρόεδρε της ΕΜΒΗ για την πρόσκληση σε αυτή τη δημόσια κρόαση με το ECDC και ευχαριστώ και τη Διευθύντρια Ανδρέα για την παρουσίαση που μας έκανε. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω δύο στοιχεία. Καταρχήν, μία συμπληρωματική ε, πρόταση στην προσέγγιση του ECDC και ε, να αναφερθώ και στο ρόλο μου ως εκπρόσωπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά το Brexit ε, κατέστησε σαφές ε, ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, δεν είναι και πολύ εξοικειωμένοι με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Και, και το ECDC έχει πρόβλημα επικοινωνίας με το ευρύ κοινό και είναι άγνωστο στον κοινό Ευρωπαίο πολίτη. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε μια πιο σφαιρική προσέγγιση. Και τα έγγραφα του ECDC υπάρχουν μόνο στα αγγλικά, δυστυχώς. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ε, διαβάζουν την ιστοσελίδα του κέντρου σας στη μητρική τους γλώσσα, κυρίως οι πιο ηλικιωμένοι που δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσετε την επικοινωνία σας με το ευρύ κοινό. Έτσι θα καταπολεμήσουμε και την παραπληροφόρηση που σοβεί σήμερα, ακόμη και για τον κορονοϊό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή και σε οργανισμούς όπως το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Όσων. Αυτό είναι σημαντικότερο και απαραίτητο περισσότερο από ποτέ στην πρόσφατη ιστορία μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους κανόνες επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής ΕΜΒ και ημών των εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECDC, εγώ εκπροσώπησα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης μαζί με την κυρία Κοπά και το κάναμε ανιδιοτελώς, αφιλοκερδί, χωρίς να λάβουμε καμία αμοιβή και θα ήθελα απλό να υπηρετήσουμε την ΕΒΗ και τους αξιότιμους ευρωβουλευτές ε, ε, χρησιμοποιώντας και μεταβάζοντάς τους τις πληροφορίες από το ECDC και δίνοντας δικές μας ε, προτάσεις. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες και ένα σύστημα feedback και αλληλοεπικοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν με καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερη επικοινωνία να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και την καλύτερη ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στους στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Κύριε Κοπά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την προλαλή σας, τη Σοφία Κούκοβιτς, γιατί είναι απολύτως απαραίτητο να εμπλέξουμε το ευρύ κοινό στη συζήτηση για θέματα υγείας. Κατά τη γνώμη μου, το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων είναι ένας οργανισμός που έχει την ικανότητα να προσαρμοστεί σε κάποιες απειλές και έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται και να αλλάζει. Το έχουμε δει επανειλημμένως και ο νέος κορονοϊός είναι μια επιπλέον περίπτωση. Ο οργανισμός αυτός έχει μια πολυσχεδή δραστηριότητα και πλευρή. Η εμπειρία μου από την τελευταία τετραετία έδειξε ότι τα δύο βασικά ζητήματα προβληματισμού είναι η μικροβιακή αντοχή και ε, ο εμβολιασμός, που είναι βασικά, δύο βασικά χαρακτηριστικά του υγειονομικού τοπίου και βασικά θέματα του κέντρου σας. Θα ήθελα επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει πιο ενεργά και να ενημερώνεται πιο τακτικά για τις εξελίξεις ε, στο έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Όσων. Και η κυρία Κουκοβίτς και εγώ ως εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπαθούμε ε, να φέρουμε κοντά το Διοικητικό Σύμβουλο στις ε, εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες ευρωεκλογές. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κοπτσίνσκα για το ενδιαφέρον που έδειξε και για την ετοιμότητά της και την προθυμία της για καλύτερη επικοινωνία πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία και με την Επιτροπή ΕΜΒΗ και με το ευρύ κοινό. Και αυτό θα είναι η σημαντική πρόκληση και για την Επιτροπή ΕΜΒΗ και για το Γραφείο Πρόληψης και Ελέγχου των Όσων. Μάλιστα. Και εσείς τι θα λέγατε κύριε Διευθυντρία. Ευχαριστώ και τις δύο εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, είχαμε επανειλημμένο στην συζήτηση αυτή στο ECDC και στο Διοικητικό Συμβούλιο και πολλά μέλη του ΔΣ δεν θέλουν άμεση επικοινωνία με το ευρύ κοινό. Θεωρούμε ότι είμαστε κάπου, με κάπου μεσάζοντες. Πάντως, σε ό,τι αφορά τη μετάφραση των εγγράφων μας, ε, όντως ε, τα περισσότερα εγγραφά μας ε, είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά. Ισχύει αυτό και το σκεφτόμαστε τουλάχιστον τις συνόψεις των εκθέσεών μας να τις μεταφράζουμε σε κάποιες γλώσσες. Γιατί τα έγγραφα που έχουμε συντάξει για τον κορονοϊό να τα μεταφράσουμε, ώστε να γίνουν μεταφράσεις έχουν αλλάξει τόσο τα στοιχεία και έχουν ε, επικαιροποιηθεί που είναι πλέον ε, απειρχιωμένα. Οπότε δεν έχει νόημα όταν είναι τόσο ραγδαίες εξελίξεις να μεταφράζουμε τα έγγραφά μας. Δεν είναι εφικτό ούτε σκόπιμο. Επίσης προσπαθούμε με, τις, με με τις μηχανικές, την αυτόματη μετάφραση, αλλά για τα τεχνικά κείμενα δεν δίνει αποτέλεσμα αυτή η αυτόματη μετάφραση. Και ευχαριστώ τις δύο εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Σοφία και τη Μαριλένα, γιατί φέρνουν τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και φέρνουν την, αυτές τις πληροφορίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECDC και το κάνουμε με πολύ καλό τρόπο. Ευχαριστώ. Ε, in weeks. Σε δύο εβδομάδες έχουμε τον Επίτροπο Υγείας. Εάν έχουμε νεότερες εξελίξεις με τον ιό αυτόν, θα καλέσουμε και εσάς για να συμμετάσχετε στην συζήτηση εκείνη. Ευχαριστούμε. Um, λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, δεν θα ψηφίσουμε σήμερα, θα ψηφίσουμε στο Στρασβούργο όταν θα έχουμε την τελική σύνθεση, τη νέα σύνθεση της Επιτροπής. Προτού πάω στην αντίρρηση, μία επίσημη ανακοίνωση για την σύσταση των συντονιστών ε, της 20 Ιανουαρίου να ελέγξω ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για τα πρακτικά της συνάντηση των συντονιστών. Ωραία. Σχετικά με τα εκχυλίσματα πρόπολης τώρα και τη σχετική αντίρρηση, παρακαλώ η κυρία Μπουινά για το ID. Αγαπητέ Πρόεδρε, επειδή συνάδελφοι, οι αντιρρήσει της Ζωέλ Μελά ε, τις παρουσιάζω εγώ γιατί δυστυχώ δεν μπορούσε... Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος διακόπτοντα. αν μπορείτε να ε, βγείτε από την αίθουσα σας παρακαλώ. Η κυρία Διευθύντρια θα, θα μπορούσα να σας ζητήσω να εξέλθετε διότι έχουμε συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρο. Ναι, Πρόεδρε, ε, παρουσιάζω λοιπόν την αντίστοιχη συναδέλφου ε, κυρίας ε, Ζουέλ Μελά που δεν μπορούσε να είναι εδώ παρούσα για να την παρουσιάσει αυτοπροσώπως. Τα πιο σημαντικά λοιπόν σημεία σχετικά με αυτήν την περίεργη απόφαση της Επιτρόπου για την ε, πρόπολη ως βασική ουσία. Είναι φυσικό προϊόν που συλλέγεται από τις μέλισσες και γνωρίζετε ότι η μέλισσα έχει επίσημα αναγνωρισμένο καθεστώς ε, ως πηγή ε, ανθρώπινης τροφής. Έχουμε επιστημονικές συστάσεις και πλαίσια που διέπουν τη συλλογή αυτή ε, είναι συμπλήρωμα διατροφής υπό και πάλι ε, αυστηρές ε, οδηγίες. Υπάρχουν σκευάσματα για τον πονόλεμο που πολλούνται με βάση εκχυλίσματα της πρόπολης. Έχει αυστηρότατα κριτήρια ασφάλειας για την ανθρώπινη κατανάλωση. Επίσης επιτρέπεται προς ανθρώπινη κατανάλωση. Είναι εγκεκριμένη δηλαδή ως ουσία αναφέρεται η Επιτροπή σε αλλεργιογόνους παράγοντες και κινδύνους και την ενδοκρινική διαταραχή και τοξικότητα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν μπορεί παρά να σκεφτεί κανείς ότι είναι φάρσα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δραστικές ουσίες των συσκευασμάτων στα οποία αναφέρεται. Γιατί να επιτρέπουμε για 10 έτη την γλυφοζάτη που είναι καρκινογόνος ε, και δεν είναι και συμπλήρωμα διατροφής όπως η πρόπολη. Η έγκριση της πρόπολης ως βασική ουσία ε, δεν αφορά παρά συγκεκριμένα φυτά τα οποία δεν είναι προς ανθρώπινη κατανάλωση σήμερα. Επίσης, είναι η δεύτερη φορά που η Επιτροπή αποκλεί την αδειοδότηση ε, ζυζανιοκτώνων χαμηλού κινδύνου. Εάν θέλουμε πραγματικά λοιπόν να έχουμε βιώσιμα εργαλεία και μέσα και λύσεις για τους γεωργούς μας, για τους καλλιεργητές, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις ε, προελεύσεις των προϊόντων αυτών. Ε, σχετικά λοιπόν με την αντίρρηση αυτή καλώ όλους τους συναδέλφους πέρα από κομματικές ή πολιτικές διαφορές να υποστηρίξουν τη θέση μας και την αντίρρηση αυτή. Θα δώσω το λόγο στις ε, πολιτικές ομάδες ξεκινώντας από το ΕΛΚ παρακαλώ. Ναι Πρόεδρε ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ε, το επιχείρημα που χρησιμοποιείται είναι ότι ε, εάν μπορούμε να χρησιμοποιούμε την πρόπολη σε σκευάσματα ε, είναι ασφαλής και για αλλού. Ωστόσο, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων που του ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει επιστημονική γνωμοδότηση για βασικές ουσίες εντός της εκθέσεως που υπέβαλε αναφέρθηκε ο οργανισμός στην γαλλική επιχείρηση που, παράγει τα σκευάσματα αυτά για σκευάσματα αντιμετώπισης των μυκητών στα φυτά. Παρότι η, έκθεση της ΕΦΣΑ δεν αναφερόταν σε άλλες απειλές ή κινδύνους, δεν αποδεικνυόταν ε, η απουσία άλλων γενετικών ή ενδοκρινικών απειλών ή στην έκθεση οι ανησυχίες που αναφέρονται στην ουσία λοιπόν δεν μπορούσαν να αποκλειστούν και κατά την άποψή μου η τεχνική και επιστημονική γνωμοδότηση πρέπει να γίνει σεβαστή. Η ουσία πρέπει να εγκρίνεται μόνο εφόσον έχουμε ε, συγκεκριμένες αποδείξεις για την απουσία ενδοκρινικής δραστηριότητας ή άλλων απειλών. Επομένως εγώ δεν υποστηρίζω την αντίρρηση. Μάλιστα. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες δεν ε, έχουμε εκπροσώπους, εκτός αν η Μισελ Ριβαζή πήγε στους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Όχι, δεν έχουμε από τους σοσιαλιστές λοιπόν. Από το κανένας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. To be forced to... Μερικέ φορές αυτή είναι η μοίρα του συντονιστή να αναγκάζεται να απαντήσει σε τέτοιου του ερωτήματα. Νομίζω ότι υπάρχει μία παρεξήγηση εδώ. Στα έγγραφα αναφέρεται με σαφήνεια ότι η πρόπολη ως φυσική ουσία θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτή, υδροδιαλυτή. Αυτό που έχουμε όμως ενώπιό μας δεν μιλάει για κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε εθανόλη που χρησιμοποιείται ως διαλυτής στο κύλισμα της πρόπολης. Οπότε δεν είναι υδροδιαλύτη η ουσία, άρα διαφορετικό ζήτημα και άρα είμαστε κατά της αντίρρησης. Μάλιστα, η πράσινη τώρα. Πάρης. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε την επιστήμη. Και αν υπάρχει υποχρέωση, επίσημη υποχρέωση εκπόνησης μελετών και μετρήσεων για να εγκριθεί μια ουσία, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί είναι φυσικής προέλευσης ή συνθετική η ουσία, αλλά να εμείνουμε στα πορίσματα των επιστημόνων. Και αν η πρόπολης ή το χείλισμα πρόπολης ή ο προμηθευτής, ο παρασκευαστής δεν μπορεί να παράσχει αυτές τις μελέτες που απαιτούνται, δεν θα λάβει και την αδειοδότηση για τη διάθεση των συσκευασμάτων του. Δεν υποστηρίζουμε λοιπόν την αντίρρηση. Από το ECR, ο κύριος Βόντρα. Ευχαριστώ. Ούτε και εμείς θα υποστηρίξουμε την αντίρρηση. Κυρίως επειδή για το εκχύλισμα της πρόπολης ε, οι πληροφορίες που είχαμε δεν ήταν αρκετές ώστε ε, να καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια για την έγκριση της πρόπολης ως βασικής ουσίας όπως προβλέπει το άρθρο 23 του κανονισμού για την φυτοπροστασία. Πάντως η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν εμποδίζει την υποβολή αιτήσεως για την ε, έγκριση του χειλίσματος πρό, πρόπολης ως δραστικής ουσίας ή χαμηλού κινδύνου βάσει του άρθρου 7 του σχετικού κανονισμού. Ω δραστική ουσία μέσου ή χαμηλού κινδύνου. Οπότε, βάσει το άρθρο 23, και επειδή δεν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 23, δεν υποστηρίζουμε την αντίρρηση. Αλλά υπάρχει μια δυνατότητα για την έγκρισή τη με άλλη μορφή στο μέλλον, γιατί εμεί αγαπούμε την πρόπολη. Κύριε κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μέλισσες είναι φανταστικά ζώα, επικονιάζουν τα λουλούδια, φτιάχνουν μέλι, βασιλικό πολτό και πρόπολη. Οι άνθρωποι επίσης ε, χρησιμοποιούν την ε, πρόπολη για να θεραπεύουν τις ε, ουλές, τις πληγές. και θα πρέπει να γίνει πιο εύκολο αυτό γιατί αν μπορούμε να την αγοράσουμε στο κατάστημα γιατί να μην μπορεί να εγκριθεί ως ε, φαρμακευτική ουσία αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτήν την διαδικασία. Το έχουμε δει και στο παρελθόν και στην Ολλανδία ε, πόσο εύκολα τα, οι λεγόμενες ε, ουσίες χαμηλής επικινδυνότητας μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνες ε, για τα ζώα και για το περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τις υπόλοιπες ουσίες που θα χρησιμοποιούν. Αν δεν γίνουν αυτές οι δοκιμές και πριν ολοκληρωθούν ε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για να αποκλειστούν ε, πιθανώς τοξικά, τοξικές παρενέργειες και χωρίς να γίνει αυτό δεν μπορούμε να εγκρίνουμε την ε, ουσία αυτή. Για τους λόγους αυτούς εμείς θα καταψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, Γενική Διεθνής Υγείας, ο κύριος Μπέρεντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι ιδιαίτερα λακωνικός γιατί μετά την συντάκτηρα της αντίρρησης. Όλοι οι υπόλοιποι ομιλητές ε, είπαν αυτά που θα ήθελα να πω κι εγώ. Η έγκριση της πρόπολης ως βασικής ουσίας, γιατί αυτό είναι το σημαντικό εδώ. Βασική ουσία είναι σημαντικός χαρακτηρισμός των δραστικών ουσιών με βάση τον κανονισμό για τη φυτοπροστασία δεν είναι χρονικά περιορισμένη και δεν απαιτείται αδειοδότηση. Μετά την έγκριση δηλαδή τα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσω για φυτοπροστασία. Γι' αυτό και τα κριτήρια του κανονισμού για την έγκριση τέτοιων ουσιών ως βασικών είναι πολύ ψηλά. Και ένα από τα κριτήρια αυτά είναι να μην είναι ανησυχητικέ. Το κύλισμα της πρόπολης με βάση τις ενδείξεις που υπέβαλε ο ίδιος ο Ετών είναι δερματικός ευαισθητοποιητής και έχει ταξινομηθεί για την ιδιότητα αυτή και άρα είναι προβληματική ουσία, είναι ανησυχητική. Δεν μπορεί λοιπόν να εγκριθεί ως βασική ουσία δυνάμει του κανονισμού. Οι άλλες χρήσεις που αναφέρονται είναι η παραδοσιακή ιατρική. Ούτε και αυτό είναι συγκρίσιμο όμως, γιατί για ε, χρήση δια του στόματος. Εδώ μιλούμε για ευαισθησία του δέρματος και μιλούμε κυρίως για φρούτα που θα ξεφλουδιστούν και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του πάνελ του ΕΦΣΑ του 2010, που κατέληξε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς πληροφορίες για να προσδιοριστεί η σύνδεση μεταξύ της κατάστασης, της κατανάλωσης της πρόπολης και των ισχυρισμών υγείας που αναφέρονταν. Οπότε, καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα με τον κύριο Βόντρα, ότι ε, η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση της πρόπολης ως βασικής ουσίας, αλλά υπάρχει δυνατότητα να εγκριθεί ως ε, δραστική ε, κανονική δραστική ουσία ή χαμηλού κινδύνου δραστική ουσία, αρκεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι γονιδιοτοξική ή ενδοκρινικός διαταράκτης. Η δεμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εγκριθεί ως δραστική ουσία. Μάλιστα, η θέση των πολιτικών ομάδων ήταν ξεκάθαρη. Θα ψηφίσουμε το Φεβρουάριο στην ΕΒΗ. 13-18 ε, πάντως το Φεβρουάριο. Και περνάμε στο συνήθι ύποπτο την αντίρρηση για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Η τηλιμέτς κανονικά είναι η πρώτη, αλλά απουσιάζει. Όχι, είναι παρούσα. Έφτασε και όλα η ώρα μου. Ναι, ήρθε η ώρα να μας παρουσιάσετε την καντήρηση. Για ακόμη μια φορά. Η παραγωγή είναι βασικός λόγος ε, της αποψήλωσης ε, σε μεγάλο βαθμό της Νοτιοαμερικής και 100% της σόγιας που καλλιεργείται εκεί είναι γενετικώς τροποποιημένη. Αυτή η μεταλλαγμένη σόγια είναι θεκτική σε ε, φυτοφάρμακα όπως η γλυφοσινάτη και η γλυφοσάτη. Οπότε ήδη τέτοια προϊόντα ψεκάζονται σε προβληματικά οικοσυστήματα, ήδη εύθραυστα. Οπότε οι μαζικέ εισαγωγέ σόγια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ζωοτροφή συμβάλλει στη μαζική καταστροφή των οικοσυστημάτων στην Νότια Αμερική. Και αν θέλουμε να πρωτοστατήσουμε στην καταπολέμηση την αποψήλωση των δασών και στην απώλεια τη βιοπικιλότητα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αμφισβητήσουμε αυτό το παράλογο σύστημα. Οπότε ρωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να συμπεριλάβει τις ε, εισαγωγέ γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων και κυρίως σόγιας ε, στην οικολογική αξιολόγηση των εισαγωγών τη, δεδομένη της ε, έλλειψης, της αποψήλωση και της, των κλιματικών, της κλιματικής έκτακτης στον έλεγχο επιπτώσεων. Γιατί, δεν, γιατί συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοδοτεί μεταλλαγμένα προϊόντα για εισαγωγέ. Αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επίγουσα ανάγκη τη μείωση τη παραγωγή και κατανάλωση ε, ε κρέατο και γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί ζητούμε να συμπεριληφθεί στη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο και μία πρόταση για τοπική παραγωγή πρωτεϊνούχων. Ευρωπαϊκή δηλαδή. Σας ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρο. Τώρα, να ακούσουμε τις πολιτικές ομάδε ξεκινάς το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εφόσον η ΕΦΣΑ, μάλλον, ότι η ΕΦΣΑ ε, έδωσε θετική γνωμοδότηση και δεν ε, διαφοροποίησε καθόλου τον, την γενετικό τροποποιημένη σόγια από την υπόλοιπη ως προς το ζήτημα που συζητούμε. Επίσης, ε, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε προηγούμενο καταψήφισης από τα κράτη-μέλη ε, γάματα φόμικρον σε αυτό το πεδίο. Πρέπει να ακολουθήσουμε και εδώ τις επιστημονικές συμβουλές και νομίζω ότι τηρώντα τι επιστημονικές συμβουλέ σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα όρια της η Επιτροπή. Μάλιστα ευχαριστώ SND. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε παρά τα όσα έχουν ήδη συμβεί να έχουμε μια πλειοψηφία. Μιλούμε για γενετικώ τροποποιημένη ισόγεια ε, Εμεί εξακολουθούμε να λέμε ότι υπάρχει υπερβολικά ευρεία χρήση ζανιοκτώνων. Είναι θέμα πολιτικής λοιπόν τοποθέτηση εδώ. Βεβαίω αυτό σημαίνει ότι δεν τίθεται ζήτημα ειδική πλειοψηφία και επίσης τον Ιανουάριο για τον ίδιο λόγο δεν ελήφθη κάποια απόφαση. Οπότε δεν μπορούμε να εγκρίνουμε κάτι το οποίο θέλει να κάνει η Κομισιόν χωρίς ειδική πλειοψηφία των ε, κρατών μελών. Γιατί έτσι μέχρι στιγμής τα όσα έχουν γίνει ε, από μας έχουν αγνοηθεί παρά το ότι η κυρία Φόντερ Λάιν μας είπε ότι προσεχώς θα λαμβάνει υπόψη την εγγρομοδότηση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για Ευχαριστώ πρόεδρε. Μιλούμε πάλι για μαγατάφο όμικρον και καλό θα ήταν να το συζητήσουμε αυτό το θέμα περαιτέρω. Αλλά πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί πιστεύω. Ε, δεν πρέπει να είμαστε συναισθηματικοί στην τοποθέτησή μας. Πρέπει να δούμε τα ωφέλη, τις απειλές, τους κινδύνους, την ανάπτυξη ενδεχομένως νέων τεχνικών ε, τεχνικών βελτίωσης ή ανάπτυξης νέων προϊόντων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς ως προς την επιστημονική κατεύθυνση που ακολουθούμε, συμβουλές που ακολουθούμε. Κάποιες χώρες, ναι, πράγματι, είναι εναντίον των γάμματα αφόμικρων. και φέρνουν αντίρρηση προς αποφάσεις της Επιτροπής λέγοντας ότι υπερβαίνει τα όρια αρμοδιότητό τη, Αλλά δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Καλό θα ήταν να είμαστε πιο επικοδομητικοί. Αν θέλαμε να ήμασταν θα αλλάζαμε το νομοθετικό πλαίσιο. Οι αναρρύθμιτες φορές ε, που έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις ε, με αυτό το δικαιολογητικό, με τον ε, με τη δικαιολογία δηλαδή του ότι η Επιτροπή υπερβαίνει την αρμοδιότητά τη, δείχνει ότι είναι λίγο αντιπαραγωγική αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Χρειαζόμαστε, εφόσον τα κράτη-μέλη το εννοούν, καλύτερη νομοθεσία. Μάλιστα. ID δεν έχουμε ομιλητή, ECR. Παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, συμφωνούμε με την Επιτροπή και κατά της αντίρρησης για δύο λόγους. έχουμε διάφορους ε, ακτιβιστές που έχουν προτείνει στην Επιτροπή να ακολουθήσει τις συμβουλές, εμείς, τις επιστημονικές δηλαδή, και εμείς το ίδιο θα κάνουμε. Διαδικαστικός τώρα, νομίζω 8 είχαμε μόνο σε αυτήν την εντολή, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά η ανησυχία αυτή δεν εδράζεται σε κριτήρια επιτροπολογίας επαρκώς. Η Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν έχει υπερβεί τις εκτελεστικές αμοροδιότητες, οι οποίε τηρούν την νομική διαδικασία του βασικού νομοθετήματος. Και επομένως, η υποβολή αντίρρησης για διαδικασία που δεν τηρεί τους κανόνες, κατά την άποψή μας υποσκάπτει, μειώνει το δημοκρατικό δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παράγωγη νομοθεσία και με βάση αυτή την αιτιολογία δεν πρέπει να υποστηρίξουμε την αντίρρηση. Μάλιστα. Η κυρία κάνει για την ε, ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο σε 6 χρόνια έχει εγκρίνει 43 διαφορετικά ψηφίσματα και τώρα πάμε για το 44ο για τους γενετικά τροπημένους ε, οργανισμούς. Και βεβαίως μαζί με αυτά πάει πακέτο η γλυφοσάτη και η γλυφοσινάτη. Η γλυφοσάτη βεβαίως είναι ε, γνωστή και η γλυφοσινάτη είναι απαγορευμένη στην Ευρώπη γιατί επηρεάζει το αναπαραγωγικό. Σας παρακαλώ λοιπόν σταματήστε από την Κομισιόν αυτές τις ε, αδειοδοτήσεις το άρθρο 6 δε παράγραφος 3 της Επιτροπολογίας ε, επίσης ε, λέει ότι έχετε την δυνατότητα να αρνηθείτε την αδειοδότηση αν δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών. Η ΔΕ Κομισιόν για το νομοθετικό της πρόγραμμα του 2020 λέει ότι θα έχει ως προτεραιότητα να δώσει ε, τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν ουσίες που εγκρίνει η Κομισιόν και μετά λέει ότι θέλει να βελτιώσει την διαδικασία της επιτροπολογίας και αυτό ακούγεται καλό αλλά μάλλον ε, ελπίζουμε να σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσετε την αδειοδότηση τέτοιων ουσιών που τελικά δεν τα θέλει κανείς ούτε καν ε, και όταν μπορούν να τα απαγορεύσουν τα κράτη-μέλη γιατί ας είμαστε ειλικρινείς τότε ε, απλά φορτώνει την δουλειά αυτή η Κομισιόν στα κράτη-μέλη και στο Κοινοβούλιο και δίνει τη δυνατότητα σε πολυεθνικές όπως η Μπάγερ και άλλες να ξεκινήσουν μακροχρόνιες διαδικασίες κατά των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να μην δίνεται ε, άδεια σε οργανισμούς οι οποίοι αντιστέκονται σε συγκεκριμένες ε, ουσίες. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε και πάλι πολύ προσεκτικά όλα τα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω, το είπαν κάποιοι βουλευτές, πως έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες και οπωσδήποτε σεβαστήκαμε τις ε, αρμοδιότητες που μας έχουν δουθεί. Και βεβαίως ε, τα κράτη-μέλη μπορεί να μην υπερψήφισαν, αλλά δεν καταψήφισαν και εισάγουν αυτές τις ε, ουσίες στην επικρατειά τους. Γιατί, Γιατί υπάρχει υψηλή ζήτηση για γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό, γιατί είναι ασφαλής αυτοί οι οργανισμοί, η ΕΦΣΑ έχει κάνει τη σχετική αξιολόγηση και δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν είναι ασφαλής ε, αυτοί οι οργανισμοί. Και βεβαίως ε, γεγονός είναι πως ε, τα κράτη-μέλη στη μόνιμη επιτροπή δεν γνωμοδοτούν, αλλά δεν καταψηφίζουν, αλλά ούτε και υπερψηφίζουν. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην εγκρίνουμε την, ε, τον οργανισμό, μια που υπάρχει θετική γνωμοδότηση. Η Κομισιόν δρά με βάση την ασφάλεια και βεβαίως δεσμευόμαστε και από τις διεθνείς συμφωνίες, αλλά είναι σαφές πως μια συγκεκριμένη πράξη η οποία επιβεβαιώνει την ασφάλεια ενός προϊόντος για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λύσει όλα τα ζητήματα στις διεθνείς συμφωνίες. Ε, πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά όχι με το να απορρίψουμε ένα συγκεκριμένο οργανισμό ο οποίος είναι ασφαλής και έχει εγκριθεί σύμφωνα με την νομοθεσία. Οπότε εισάγουμε επίσης, θα ήθελα να πω, ναι, από την Νότια Αμερική αλλά και από τη ΣΥΠΑ και από τον Καναδά. Περνόμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί για το θέμα της αποδάσωσης που είναι πάρα πολύ σοβαρό και γνωρίζουμε όλοι πως ε, η Κομισιόν έχει προτείνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για το θέμα της αποδάσωσης. Πρέπει να μας απασχολήσει αυτό, αλλά σας παρακαλώ όχι με το να απορρίπτουμε έναν οργανισμό που μπορεί να εισαχθεί από οποιαδήποτε τρίτη χώρα και δεν καλλιεργείται ε, απαραίτητο σε μια αποδασωμένη περιοχή. Πρέπει να είμαστε λοιπόν αποτελεσματικοί. Γιατί ε, με το να απορρίψουμε μια τέτοια ουσία ε, παρανομούμε και δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί. Οπότε να σα πω ότι δεν υπάρχει κάποιος ε, λόγος νομικός να απορρίψουμε την αδειοδότηση αυτή. Με συγχωρείτε αν ακούγομαι βαρετή, έτσι πρέπει να είναι, γιατί αυτά είναι τα νομικά επιχειρήματα. Και τονίζοντας βεβαίως ότι σεβόμαστε πλήρως τις διεθνείς ε, δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίρνουμε πολύ σοβαρά. Δεν είναι λοιπόν ε, αυτό το οποίο κάτι πρέπει να γίνει μέσω τη αδειοδότηση ενό οργανισμού. Ξέρετε ότι έχουμε σεβαστεί το δικαίωμα τη εξέταση ε, και τι σχετικέ αρμοδιότητε που υπάρχουν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε θα ψηφίσουμε στις 13 Φεβρουαρίου και αν ε, περάσει θα πάει στην Ολομέλεια. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στο Στρασβούργο, 13 Φεβρουαρίου. Λύεται η σημερινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.